Okay, colleagues, can I call the meeting to order? Αρχίζει η συνεδρία, συνάδελφοι, λέω ο πρόεδρος ο κύριος Σίμψον και θα αρχίσω ζητώντας σας την έγκριση του σχεδίου της συνεδρίας διατάξεως. Συμφωνείτε? Ε, τότε πάμε στην έγκριση των πρακτικών. Έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό? Το σημείο? Όχι. Υπέροχο. Επόμενο. Είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Βελγική Προεδρία όσον αφορά τα θέματα μεταφορών. Ο υπουργό κύριος Σου είναι εδώ και του δίνουμε τη σκητάλη. Ευχαριστώ πρόεδρε στα αγγλικά. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζει τα Ολλανδικά. Κύριοι βουλευτέ, μέλη τη Επιτροπή τη Μεταφορά στι 13 Ιουλίου του 2010 παρουσίασα τι προτεραιότητες μα για κινητικότητα και μεταφορές. Και όταν έγινε η παρουσίαση το δεχθήκατε ευνοϊκά. Βέβαια ορισμένοι βουλευτές ε, το είχαν όρισαν αυτό το πρόγραμμα ως ιδιαίτερα φιλόδοξο. Η υλοποίηση αυτών των στόχων θα είχε θα, άμα πραγματικά είχε επιτευχθεί θα σημαίνει επιτυχία της Προεδρίας. Τώρα η Προεδρία μας τελείωσε και μας είπαν ότι η Προεδρία μας έχει αποτιμηθεί θετικά για τις μεταφορές και την κινητικότητα. Σας ανέφερα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές και το Συμβούλιο Μεταφορών στην Αμβέρσα. Σήμερα θέλω να σας δώσω μια γενική εικόνα των διαφόρων αποτελεσμάτων και προόδων σε ορισμένους τομείς. Εμείς θελήσαμε να, να θελήσαμε την ασφάλεια, την ασφάλεια ως κλειδί όλων των μεταφορών κατά τη Βελγική Προεδρία. και το πρόγραμμά μας είχε προβλέψει 13 μεγάλες εκδηλώσεις που θα βοηθούσαν να προωθηθεί το θέμα της ασφάλειας. Για την αηφορία των μεταφορών. Εμείς μιλήσαμε τον Οκτώβριο σχετικά και η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν η παρουσίαση της Λευκής Βίμπλου σχετικά με την ε, στρατηγική πρόβλεψη για τις μεταφορές. Τι προσανατολισμό να δώσουμε εμείς ε, τις μεταφορές, εγγυόμενη την αηφορία και την ασφάλεια. Η Λευκή Βίβλος ε, καθυστέρησε. Αλλά εμείς δεν σταματήσαμε περιμένοντας τη Λευκή Βίβλο. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση στο Συμβούλιο για τα βασικά στοιχεία της Λευκής Βίβλου. Το αποτέλεσμα όλες αυτής της συζήτησης οδήγησε σε έναν περαιτέρω προσανατολισμό της Κομισιόν για τη σύνταξη αυτής της Λευκής Βίβλου. η οποία θα δημοσιευθεί υπό Ουγγρικής Προεδρία. Τον Οκτώβριο παρουσιάσαμε την οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου χωρίς σύνορα. Το πρώτο δηλαδή πακέτο για τους σιδηροδρόμους. Η πρώτη ομάδα για τις ε, χερσαίες μεταφορές στο Συμβούλιο ξεκίνησε την ανάλυση του σχεδίου και διαχώρισε το σχέδιο σε τρεις βασικές θεματικές για να διευκολύνει τις συζητήσεις μέσα στην ομάδα εργασίας. Οι τρεις επιλογές είναι η χρηματοδότηση και δασμολόγηση των υπηρεσιών, ρυθμιστική επαγρύπνηση και εποπτεία. Το πρώτο θέμα βελτιώθηκε μετά από κοινή συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια πρώτη επαφή για να καταλήξουμε στο συμβιβασμό στο Συμβούλιο Μεταφορών το 2010 οργανώθηκε μία συζήτηση για την επεξεργασία μίας μελλοντικής πολιτικής και να ξεκινήσουμε τις εργασίες της ομάδας εργασίας για να καταλήξει στο πρώτο εξάμεινο του 2011 σε συμφωνία πάντα υπό Ουγγρική Προεδρία. Ελπίζουμε κάτι τέτοιο να γίνει στις 16 Ιουλίου. 16 Ιουνίου διορθώνει το μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, είμαι πεπισμένος ότι η κινητικότητα στην Ευρώπη θα πρέπει να συνδέεται με την μεγαλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος. Όλα τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να γίνουν πιο οικολογικά και πιο Οικονομικά. Καταλήξαμε στην συμφωνία για την Ευρωβινιέτα, για το Ευρωσήμα. Και αυτό για να διεθνοποιήσουμε το κόστος των μεταφορών, των, των εσωτερικών μεταφορών ε, στο δρόμο. Δηλαδή, να θεσμοποιήσουμε πλέον την αρχή του ποιος ρηπαίνει πληρώνει. Δηλαδή, η Ευρωβινιέτα προβλέπει το σκέλος χρηματοδότησης των υποδομών, αλλά και την καταπολέμηση της ρήπαρσης, όπως επίσης μέσα από την Ευρωβινιέτα αποφεύγονται τα μποτιλιαρίσματα και γίνεται σεβαστός παράλληλα ο ανταγωνισμός. Όλο αυτό το ντοσιέ έχει περάσει στην Ουγγρική Προεδρία που ελπίζομαι να εγκριθεί. Για την αηφόρο κινητικότητα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αφορά και στην προστασία των καταναλωτών. Με ιδιαίτερη προσοχή στους ε, για τα άτομα με μειωμένες κινητικές δυνατότητες. Το Συμβούλιο μετά από συνδιαλλαγή με το Κοινοβούλιο κατέληξε στην προστασία των επιβατών, των λεωφορείων, αστικών και τουριστικών δηλαδή τι γίνεται σε περίπτωση δυστυχήματος, πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των αναπήρων, τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης, τι γίνεται σε περίπτωση προσφυγών. Όλα αυτά τα μέτρα θα αρχίσουν να ισχύουν για τα ταξίδια με λεωφορείο πάνω από 250 χιλιόμετρα και για τις διαδρομές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται και ένα βασικό πακέτο για τα πιο σύντομα ταξίδια και βασιζόμαστε εδώ στην προστασία των δικαιωμάτων των αναπήρων. Έχουμε μία χάρτα για την προστασία των δικαιωμάτων του επιβάτη για όλα τα μέσα μεταφοράς. Και αυτή η χάρτα θα αλλάζει ανάλογα και με την συσσωρευμένη εμπειρία. Εμείς θελήσαμε να ενισχύσουμε και το καμποτάζ, πάντα μέσα στο πλαίσιο της αηφορίας. Το καμποτάζ αφορά στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στην Ευρώπη μεταξύ ευρωπαϊκών λιμένων ή ευρωπαϊκών λιμένων και έξω λιμένων. Στις 16 λοιπόν Σεπτεμβρίου του 2010 συναντηθήκαμε άτυπα στην Αμβέρσα για τις θαλάσσιες μεταφορές. Στις 2 Δεκεμβρίου του 2010 καταλήξαμε στα συμπεράσματα και αποφασίσαμε να φτιάξουμε την Blue Belt, δηλαδή την κιανή οδό, ε, ζώνη και τις ε, κιανές διαδρομές. Δηλαδή, τα πλοία που χρησιμοποιούνται για το καμποτάζ, άσχετα από τη σημαία που φέρουν, μπορούν να έχουν αυτήν την ε, γαλάζια ζώνη ή το σήμα των γαλάζιων δρόμων. Πριν αποφασίσουμε οριστικά για την πλήρη υλοποίηση της ιδέας για τη γαλάζια ζώνη, ξεκινήσαμε στις 30 Νοεμβρίου του 2010 το πείραμα, που αποτελεί και το βασικό βήμα για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των θαλασσίων μεταφορών. Τώρα, επειδή η ομάδα για τις θαλάσσιες μεταφορές υπό Ουγγρική, Προεδρία θα συνεχίσει να προεδρεύεται από τους Βέλγους θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτά τα μέτρα. Για τις αερομεταφορές καταλήξαμε σε μια συμφωνία για τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με ένα σχέδιο δράσης που φτάνει μέχρι το 2050 και αφορά στις 150 χώρες που συμμετέχουν στη ΙΑΤΑ. Με την έγκριση αυτής της πρώτης παγκόσμιας και τομεακής συμφωνίας, οι αρχές της πολιτικής αεροπορίας κατέδειξαν ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τις κλιματικές αλλαγές. Ασφάλεια των μεταφορών. Κυρίες και κύριοι, κατά την Προεδρία μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε ένα ανακοινοθέν για τους προσανατολισμούς σχετικά με την ασφάλεια στις μεταφορές. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου που προτάθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου για να μπορέσουμε να προθίσουμε πιο σίγουρες μεταφορές. Μεταξύ των άλλων το Συμβούλιο υποστήριξε και την άποψη για την μηδενική ανασφάλεια. Κάθε θάνατος ε, ε, στις μεταφορές είναι ένας άχρηστος θάνατος και ζήτησε η Κομισιόν να εξετάσουμε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και την αηφορία. Έγινε μία συμφωνία για τη διαχείριση της διασυνοριακής κίνησης, όπου ανταλλάσσουμε ηλεκτρονικά στοιχεία για τις ε, παραβάσεις βασισμένη στο Μητρό των πλακών των αυτοκινήτων και διαπιστώνεται ο παραβάτης. Στα τέλη του χρο... της χρονιάς θα έχουμε μια νέα οδηγία σχετικά. Στις 26-28 Οκτωβρίου του 2010 οργανώσαμε μια διάσκεψη κορυφής για τις αερομεταφορές και καταλήξαμε στη δήλωση της Μπρουζ. Έχουμε εκεί πολλές συστάσεις. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αερομεταφορών της Ευρώπης, εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού με την εφαρμογή των ΦΑΠ, συστάσεις για την ασφάλεια και την ανάγκη να εγγυθούμε την αηφορία των αερομεταφορών στις αρχές Δεκεμβρίου, στο τελευταίο Συμβούλιο Μεταφοράς, αποφασίσαμε να συστήσουμε μια ομάδα εργασίας τεχνικών και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα πρέπει να βοηθήσουν τον κύριο Κάλλας και την Βελγική Προεδρία για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας της Μπρούζου. Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να αναλύσει την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας στους διάφορους τομείς των ευρωπαϊκών μεταφορών και να ελέγχει και το σύστημα ανταλλαγής των ποσοστώσεων εκπομπών. Και πρέπει να σας πω ότι μία τρομοκρατική ενέργεια σε ένα εμπορικό αεροπλάνο αποφεύχθηκε. Αλλά μετά από αυτήν την αποτυχημένη απόπειρα εμείς θελήσαμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια, τη βελτίωση των κανόνων στις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και σε δεύτερη φάση καλύτερο συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων μέσω των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων για την ασφάλεια των ΕΙΣΤΗ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε και τον τροποποιημένο κανονισμό για την εφαρμογή του MSA. Το Συμβούλιο Μεταφορών προχώρησε στην έγκριση του τρίτου πακέτου και ανέθεσε στο ΕΜΣΑ νέες αρμοδιότητες. Το Βέλγιο λοιπόν συνεχίζει να εργάζεται δυναμικά για αυτό το ντοσιέ. Πόσο μάλλον που θα συνεχίσουμε να προεδρεύουμε να συμπροεδρεύουμε μάλλον, είπαμε την Επιτροπή των Θαλασσίων Μεταφορών μαζί με τους Ούγγρους. Θα ήθελα τώρα να ολοκληρώσω αναφερόμενο στον Γαλιλαίο. Σε συνεργασία με τους Ισπανούς και την Κομισιόν καταλήξαμε σε συμφωνία για το ρόλο που θα πρέπει να παίξει ο μελλοντικός οργανισμός GNSS δηλαδή το ευρωπαϊκό GPS κυρίως για τα θέματα ασφάλειας. Ο κανονισμός 912 του 2010 δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκάτου του 2010 και από τον Νοέμβριο θα αρχίσει να ισχύει. Δηλαδή, θα αρχίσει να εφαρμόζεται το σύστημα GNSS και θα υπάρξουν όμως αλλαγές στα θέματα διαχείρισης όταν θα γίνει η αποτίμηση της λειτουργίας του συστήματος όπου θα εξετάσουμε θέματα χρηματοδότησης, ε, θέματα αποδοτικότητας κλπ. Αυτό το θέμα όμως δεν εξετάστηκε η Βελγική Προεδρία. Θα το εξετάσει η Ουγγρική Προεδρία. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο θετικός απολογισμός δεν είναι καρπός των εργασιών του Προέδρου, του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, είναι καρπός ε, της συνεργασίας όλων των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συμμετοχή και την υποστήριξη στο έργο της Βελγικής Προεδρίας. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για την οδηγία Cross Border, την Ευρωβινιέτα και επίσης για το MSA και όλα τα θέματα των αερομεταφορών. Ήταν μεγάλη μου χαρά που μπόρεσα να εργαστώ μαζί σας για να προχωρήσουμε όλα αυτά τα ντοσιέ χέρι με χέρι. Σας ευχαριστώ. Thank you, uh, Minister. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πέντε από τους συντονιστές έχουν ζητήσει το λόγο. Ας δώσουμε τρία λεπτά στον καθέναν για να μπορέσουν να μιλήσουν και άλλοι. Ο κύριος Γκρός πρώτα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εξ ονόματος του ΕΛΚ και όλων των συναδέλφων, όχι μόνο όσων είναι εδώ, αλλά και των υπολείπων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και εσάς και τους ε, συναδέλφους σας και, τον, ε, και τη μόνιμη αντιπροσωπεία. Δεν έχουμε απλώ αγαστή συνεργασία, αλλά έχουμε και συνεργασία σε ό,τι αφορά την εμπειρογνωμοσύνη. Και αυτό είναι πάντα καλό γιατί οδηγεί σε σωστέ αποφάσει. Εσεί Είχατε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα και κρατήσατε το λόγο σας που δυστυχώς δεν συμβαίνει πολλές φορές στην πολιτική. Αλλά νομίζω ότι από τον Δεκέμβριο του 2008 ήταν αυτός ο φάκελος στο Συμβούλιο και αφορούσε πολύ, σημαντικές, πολύ σημαντικά θέματα όπως την διασυνοριακή ποινική δίωξη, την Ευρωβινιέτα που πήγε το 2009 στο Συμβούλιο και πάλι δεν κινήθηκαν πάρα πολλά ως προς αυτό, τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Είχαμε, παρα, είχαμε ξεχάσει ότι θα μπορούσε να υπάρξει ελπίδα, είχαμε ξεχάσει ότι θα μπορούσε να καταλήξει κάπου όλη αυτή η υπόθεση, αλλά τελικά τώρα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Είχαμε αποκαρδιωθεί. Οι προσεγγίσεις σας λοιπόν και οι προσπάθειές σας όντως βοήθησαν. Πολλές φορές το Κοινοβούλιο αμφισβήτησε το αν θα υπάρξει πρόοδος, αλλά νομίζω ότι αυτά τα τρία παραδείγματα ήταν πάρα πολύ σαφή και πρόδειλα της προθέσεώς σας να προχωρήσετε, ειδικά σε ό,τι αφορά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου γιατί συνήθω τα κράτη-μέρη παίρνουν πολύ εθνικέ αποφάσει και όχι τόσο πολύ ευρωπαϊκέ. Έχουμε λοιπόν δείγματα για την διασυνοριακή συνεργασία, για την βιωσιμότητα τη πολιτική και σε ό,τι αφορά του ε, ε, ταξιδιώτε. Του επιβάτε και τα δικαιώματά τους και αυτό θα είναι σημαντικό όχι μόνο για τώρα αλλά και για το μέλλον, γιατί μετά θα υπάρξει και το συνολικό πακέτο το οποίο πρέπει να δούμε, έτσι ώστε να είναι πιο διαφανέ, πιο απλό για του πολίτε και να μην δημιουργεί αιτίε για παράπονα και προβλήματα στου ε, επιβάτε. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε στο, στο μέλλον. Η Ευρωβινιέτα, εντάξει, κατάληξαμε σε ένα συμβιβασμό. Οι συμβιβασμοί πάντα είναι δύσκολοι, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι, αλλά νομίζω ότι έχουμε διατηρήσει έναν τύπο του earmarking ε, δεν χρειάζεται να είναι υποχρεωτικό, αλλά οι, ε, οι δαπάνες που, οι ε, επενδύσεις που μπορούν να έρθουν από τον τομέα των, ε, ε των μεταφορών, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η χρηματοδότηση. Αυτό το κάνουμε, πρέπει να το δούμε μάλλον όχι μόνο στις, επενδύσεις αλλά και σε, άλλα, σε άλλους τομείς. Ε, Διευθυντικά ταμεία α πούμε που πάντα δίδονται μεγάλα ε, ποσά και ποτέ δεν γίνονται συζητήσεις για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε εμείς στον τομέα των μεταφορών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που κερδίσατε εσείς, τον πόνους που κερδίσατε από το Συμβούλιο με τις αποφάσεις σας θα μπορέσει νομίζω να προχωρήσει το θέμα της χρηματοδότησης και σε άλλους, ε, και σε άλλους τομείς. Και επίσης η ασφάλεια κύριε Πρόεδρε. Μιλώ για τις ε, αεροπορικές μεταφορές. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητα από τα θέματα που συζητούμε εδώ μαζί σαφές, σαφείς γνωμοδοτήσεις και στο Συμβούλιο Μεταφορών για συγκεκριμένα θέματα. Ας πούμε συνέπειες ε, του ηφαιστείου και της τάχτης που ζήσαμε ε, έγιναν άμεσες παρεμβάσεις τότε, ίσως λίγο, πολύ γρήγορες, αλλά αυτό που λείπει είναι να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα από αυτές τις δράσεις και από αυτές τις, από αυτές τις φυσικές καταστροφές που πολλές φορές συμβαίνουν και να μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα. Φυσικά είναι σημαντικό να υπάρξει έλεγχος και στο συνολικό σύστημα, αλλά αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι χρειάζεται σαφής ε, ε, ένδειξη για ε, επίτευξη πρόοδου. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τις προσπάθειές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά αποτελέσματα στα οποία καταλήξατε. Ευχαριστώ. Ε, πολύ έτσι, γενναιόδωρα τα τρία λεπτά που σας δώσαμε νομίζω. Καλύτερα να μείνετε στα τρία λεπτά. Τρία λεπτά είπαμε. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα συμφωνήσω γενικώ με αυτά που είπε ο συνάδελφός μου, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και την ομάδα σας ε, και όλους τους μόνιμους προσώπους για την εξαιρετική εργασία που έκαναν Πραγματικά ήταν πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα και χαίρομαι που επιτύχαμε ένα μεγάλο τμήμα αυτού. Έχουμε τη Λευκή Βίβλο. Εκεί υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Ε, μιλούμε όμως για ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό όραμα για την, ε, για την πολιτική, για την κινητικότητα και τι μεταφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα ήθελα να είχε γίνει πραγματικότητα κατά τη διάρκεια τη Βελγικής Προεδρία. υπήρξαν κάποιε καθυστερήσεις, δεν τα καταφέραμε. Αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικέ συζητήσει ω προ αυτό, ειδικά για το, για το μέλλον των μεταφορών των σιδηροδρομικών. Έγιναν κάποιε αναφορέ και στην αναθεώρηση του πρώτου πακέτου για του σιδηροδρόμους. Υπάρχουν όμω και άλλε πτυχέ που πρέπει να δούμε από κοινού με αυτό, α πούμε οι πηγέ χρηματοδότησης ε, για τι υποδομέ επίση και η διαλειτουργικότητα που πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεκριμένη και να είναι και πιο απτή μεταξύ όλων των τομέων ε, ε, μεταφορών. Αυτά τα θέματα είναι πολύ πιεστικά και πρέπει να τα δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το συντομότερο δυνατόν. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρόνο που δόθηκε στα διάφορα ζητήματα στο Συμβούλιο και τα θέματα που αφορούν κυρίως το φάκελο και τις μεταφορές, με δεδομένο ότι ήταν πολύ σφιχτό, πολύ αυστηρό το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το ότι επιτεύθηκαν όλα αυτά τα σημαντικά. Συνήθω ε, είναι δύσκολο να επιτύχουμε πλειοψηφία για τέτοιου σημαντικού φακέλους και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο πολλές φορές να καταφέρουμε τελικά να έχουμε κάτι ε, φιλόδοξο στον τομέα των ε, μεταφορών. Αναφέρατε το φάκελο για την με την Ευρωβινιέτα. Πολύ σημαντικό και πολύ σωστό που λήφθη υπόψη η άποψη του Συμβουλίου. Βεβαίω δεν έχουμε φτάσει στο τέλο όλη αυτή τη ιστορία ακόμη και σε ένα βαθμό ξέρετε ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Ευελπιστώ ότι σε αυτό το ζήτημα, καθώς επίσης και στους ε, παραβιάσεις που γίνονται από διάφορους μεταφορείς, ε, εσείς ως μέλος του Συμβουλίου θα συνεχίζετε να πιέζετε έτσι ώστε να δούμε το θέμα αυτό από την ευρωπαϊκή του πλευρά και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Ε, αναφέρατε και κάποιες, ε, κάποια θέματα που αφορούν τις αεροπορικές μεταφορές, τις ε, θαλάσσιες μεταφορές, την ΕΜΣΑ, τον ενιαίο ουρανό, το 2012. Το... Ελπίζω ότι το Βέλγιο θα συνεχίσει να πιέζει για να προωθηθούν όλοι αυτοί οι φάκελοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πραγματικό χώρο ευρωπαϊκών μεταφορών και κλείνοντα, Πρόεδρε, για τα δικαιώματα των επιβατών, φυσικά αυτό είναι μια επιτευθύνσα συμφωνία, δεν είναι ιδεατή, όλοι έπρεπε να κάνουμε κάποιου συμβιβασμού, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ένα βήμα προς τα μπρος. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών και ειδικά στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Περιμένουμε βεβαίως και την πρωτοβουλία ίσως που θα υπάρξει από την Κομισιόν. Κλείνοντας λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, προσπάθειές σας, για τη βοήθειά σας και για τη συμβολή σας. Εγώ θα ε, ελπίζω ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε να πιέζετε. Η κυρία Μάισνερ από τους φιλελεύθερους. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ. Θα ήθελα να διαφοροποιηθώ λίγο από τους προηγούμενους. Καταρχάς να πω τι είναι αξιόλογο από τη δική μου την ε, πλευρά. Ε, όταν ξεκίνησε η Βελική Προεδρία δεν ξέραμε καν αν θα υπάρξει αλλαγή κυβέρνηση ή όχι. Υπήρξαν κάποιοι φόβοι ότι θα μπορούσαν να καταρρεύσουν οι εργασίε τη ε, Προεδρία. Χαίρομαι που όλα πήγαν καλά, που δεν είχαμε τέτοιε καταστροφέ. Που, ε, βέβαια εντάξει, δεν είχατε νέα κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι καλό. Το γεγονό ότι δεν έχουμε καθόλου κυβέρνηση βέβαια είναι άλλο θέμα τώρα για τα δικαιώματα των επιβατών, νομίζω ότι το, ε, έτσι όπως ε, το ε, διαχειρίστηκε η Προεδρία, ε, εντάξει, δεν, η Προεδρία μπορεί να επιτύχει μόνο όσα της επιτρέψουν τα κράτη-μέλη να επιτύχει. Οπότε είναι ε, είναι λυπηρό που έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι καλό που υπάρχει βέβαια το όριο αυτό των 250 ε, ε, χιλιόμετρων, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό δεν βοηθά πάρα πολύ τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Εντάξει, όλα είναι, είναι διαδικασίε που, πολιτικέ που δεν μπορούμε και σαφώ να επηρεάσουμε. Ευρωβινιέτα, βεβαίω, μπράβο σα. Αυτό τώρα που υπάρχει ε, ε, στο τραπέζι από την ε, Προεδρία είναι λίγο, γιατί σημαίνει ότι θα υπάρξουν περισσότεροι φόροι, αλλά τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Και ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τους, Ουγγαρ, με τους Ούγγρους. Γιατί ε, θεωρούσαμε ότι ε, σας εμπιστευόμασταν μάλλον εσάς περισσότερο, να πετύχετε περισσότερο. Ίσως ε, με την ε, Προεδρία αυτό να είναι λίγο πιο δύσκολο. πρέπει να, περιμέναμε περισσότερο, είναι αλήθεια αυτό. βέβαια υπήρξαν κάποιες προτεραιότητες οι οποίες τέθηκαν από τη δική σας, από τη δική σας Προεδρία. ειδικά τα αποτελέσματα για τις αεροπορικές μεταφορές ήταν καλά και μπράβο σας. Επίσης το θέμα της, ε, των ε, αεροπορικών, ε, των τρομοκρατικών επιθέσεων σε, με αεροπορικά μέσα ήταν πολύ σημαντικό που το θίξατε. Γενικώ πώς λοιπόν υπάρχουν πολλά θετικά σημεία, υπάρχουν πολλά σημεία για να σας επενέσει κανείς, αλλά υπάρχουν και δύο-τρία πραγματάκια τα οποία ήταν λίγο απογοητευτικά που ήθελα έτσι να σας τα αναφέρω εξ ονόματος της ε, ομάδος μου. Ελπίζω να κράτησα το όριο των τριών λεπτών, Πρόεδρε. Ναι, ναι, το κράτησες. Ευχαριστώ. Η πράσινη, ο κύριος Κράμερ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, δύο πράγματα αναφέρατε. Τα κλείσατε. Ένα η Ευρωβινιέτα και ένα τα δικαιώματα των επιβατών η Ευρωβινιέτα, το, ότι, το γεγονός ότι την ξεκινήσατε και ότι φτάσατε σε ένα αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό γιατί πριν από, πριν από σας δύο προεδρίες το προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Αλλά η Ευρωβινιέτα δεν νομίζω ότι είναι ένας επιπλέον φόρος. Η Ευρωβινιέτα έχει, ε, έχει κάνει μια πρόοδο, έχει οδηγήσει μια πρόοδο, γιατί μιλάει για εσυντορήκευση των εξωτερικών, του εξωτερικού κόστους. Μιλούμε για ε, δίκαιο ανταγωνισμό σε, ε, σε, σε τομείς, που ουσιαστικά, τομείς μεταφορών που ουσιαστικά απέχουν χιλιόμετρα ο ένας από τον άλλον. Γιατί ισχύει για όλους τους δρόμους, για όλα τα οχήματα, μιλάτε για διόδια, τα οποία αν θα αρθούν είναι θέμα των κρατών μελών. διόδια ας πούμε πολύ ψηλά όπως, όπως υπάρχουν στην, ε, ε, στην ε, Ελβετία. Είναι πολύ άδικο. Και αν λέτε τώρα εσείς ότι, είσαστε, ότι η Ευρωβινιέτα είναι ένας, ένας επιπλέον φόρος, εγώ δεν συμφωνώ. Όλα αυτά τα έχουμε δει και σε ό,τι αφορά τις, και, και άλλους τομείς μεταφορών. Εμείς υποστηρίζουμε τη φορολογική πολιτική των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χωρίς Χωρί συγκεκριμένα μέτρα δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και σε άλλους τομείς όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές οι οποίες επίσης επηρεάζονται τραγικά από τι μεταφορές Δικαιώματα των επιβατών. Ήσασταν πάρα πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά τους ε, σιδηροδρόμους. Τώρα έχουμε 250 ε, χιλιόμετρα για τα, ε, για τα λεωφορεία, 5 ώρες έχουμε για τα αεροπλάνα, το δικαστήριο είπε αποκλείεται να γίνει αυτό, 3 ώρες κάντε το. εν πάση περιπτώσει όμως, αν το αεροπλάνο έρθει, έρθει στην ώρα του, καλά. Αν δεν έρθει όμως όλοι συνέχεια μας λένε εντάξει θα έρθει, περιμένετε 10 λεπτά, περιμένετε 10 λεπτά και καταλαβαίνετε ότι ξεπερνάμε το όριο που έχουμε θέσει. Γιατί όμως είναι τα, οι ενδιάμεσες πτήσει, α πούμε και, το, και η ώρα που περιμένει κανείς γιατί είναι τόσο σύντομη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ε, το δούμε το θέμα και να επιβάλλουμε πολύ πιο αυστηρού κανόνε. Ξέρω ότι έχετε ε, επιτύχει καλά, ξέρω ότι για την Ευρωβινιέτα ήταν σημαντικό ο συμβιβασμό στον οποίο καταλήξατε. Οπότε συνεχίστε και τώρα ως απλό κράτος μέλος να πιέζετε για να έχουμε πιο δίκαιο ανταγωνισμό γιατί όντως πρέπει να προωθήσουμε τις, ε, τους φιλικούς προς το περιβάλλον τομείς μεταφορών. Κλείνω, Πρόεδρε, και να πω ότι μιλήσατε για την ευελγική ευρωβινιέτα. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς ακριβώς εφαρμόζεται η Ευρωβινιέτα ε, όπως, για να μην γίνει όπως αυτό στην, ε, όπως στην Ολλανδία που είπαμε εντάξει ε, συμφωνούμε σε κάτι αλλά τελικά εξαφανίστηκε. Το βελγικό δίκαιο είναι συμβατό με, την, με, την, με το ευρωπαϊκό δίκαιο ώστε να μην φορολογούνται μόνο οι αλλοδαποί. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς ακριβώς εφαρμόζεται η βελγική Ευρωβινιέτα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντάλ. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, eh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ, Πρόεδρε, για τα όσα επιτύχατε κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας. Χαίρομαι πολύ που βάλατε τις ιστορικές μεταφορές στην ατζέντα. Εδώ, εδώ, στα δεξιά είμαι, εδώ, από εδώ, στα δεξιά. Και όπως σας έλεγα, με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι στην ατζέντα έχετε βάλει και τα θέματα των μεταφορών. Και θα γνωρίζετε για το Ρήνο ότι ο Ρήνος έχει μπλοκαριστεί διότι έχει βυθιστεί κάποιο σκάφος. Και έχουμε άλλα 200 περίπου σκάφη τα οποία έχουν μπλοκαριστεί η παραγωγή σταμάτησε, όλη η οικονομία έχει θυγεί. Υπάρχει επομένω εδώ ένα πραγματικό πρόβλημα. Βέβαια γνωρίζω ότι ακόμη ασχολείστε με την ομάδα εργασία για τα θέματα μεταφορών και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε ε, αν μπορείτε και αυτό να το βάλετε στην ε, ε, ημέρησια διάταξη. Μιλάμε για το Ρήνο, δεν λέμε για κάπου στη μέση του πουθενά. Επομένως, εμείς υπολογίζουμε στο ενδιαφέρον σας. Επίση, μια που θα συνεχίσετε να ασχείτε την Προεδρία της ομάδα για τις μεταφορές στον ε, Διεθνή Οργανισμό για τη Θάλασσα, ε, τι θα γίνει με αυτές τις ποσοστώσει που προβλέπουν όσον αφορά την ε, Βαλτική. Στον ΆΕΜΟ, επομένως, παρακαλώ, βάλτε και αυτό το θέμα προ συζήτηση. Τι γίνεται με αυτή την μπλε γαλάζια Ευρώπη που θέλουν να πετύχουν. Θέλουν για όλη την Ευρώπη να ισχύουν αυτά τα μέτρα, βαλτική κλπ. Θέλησαν πάρα πολύ θετικό το ότι μας μιλήσατε για τρόπους μεταφοράς φιλικούς προς το περιβάλλον και στις πρωτές οδούς, όχι μόνο για το σιδηρόδρομο και τα, τις μεταφορές. Όπως ξέρετε στις κατοχώρες έχουν μια νέα κυβέρνηση και αποφάσισαν να μην προωθήσουν καθόλου αυτό το μέτρο το οποίο συζητεί σε επίπεδο Ευρώπη. Πρόεδρο, ο κύριο Στέρξ έχει ζητήσει το λόγο. Αν δεν ζητήσει άλλο το λόγο, σε μιλήσει τώρα ο κύριο Στέρξ και εδώ ο υπουργό σα απαντήσει όλου. Εντάξει, δεν έχει το λόγο. Ναι, πρόεδρε. Κρίμα που δεν είχαμε την άνοιξη πέρσι, την λευκή βίβλο όπως θελήσαμε. Θα μπορούσαμε, αν υπήρχε λευκή βίβλος, να αρχίσουμε την συζήτηση. Κρίμα. Έτσι θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε τι θα γίνει όπως το 2020. Πάντως νομίζω ότι για κάποια μέτωπα έχουμε ε, καταφέρει κάποια πρόοδο. Ιδίως όσον αφορά το earmarking και γι' αυτό και τα κράτη-μέλη. Δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένο. Γιατί τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί με το earmarking είναι γνωστά. Αλλά δεν αρέσουν πάρα πολύ στα κράτη-μέλη αυτά που ανακοινωθεί. Μιλάμε για εσωτερήκευση, μιλάμε για το κόστος του εξυγχρονισμού, για την υποδομή γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε εξαφάνιση του εξωτερικού κόστους. Εμείς ελπίζουμε όντω να μην μηδενιστεί Αλλά δεν είναι λογικό κανείς να προσπαθεί να μειώσει το εξωτερικό κόστος με οποιαδήποτε θυσία. Θέλω να συμφωνήσουμε εμεί εδώ και α ε, πείσουμε τους συναδέλφους που δουλεύουν σε άλλες επιτροπές. Τώρα, όσον αφορά την, ε, την πολιτική μεταφορών, όταν έρχεται η ώρα να έχουμε επαφές με το Συμβούλιο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί τα περισσότερα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι θέμα εθνικής πολιτικής και είναι δύσκολο, επομένως, να έχουμε διασυνοριακή πολιτική και ρυθμίσεις. Άρα να δούμε κατά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο και έτσι να ωφεληθούν και οι εμπορευματικές μεταφορές αλλά και η μεταφορά πιβατών. Άκουσα τον συνάδελφο Κράμερ. Ότι δηλαδή πρόκειται για το σιδηρόδρομο, ο οποίος είναι το θεμέλιο, η αφετηρία για τις μεταφορές, αλλά αυτά τα λέμε πάρα πολλά χρόνια. Και όσον αφορά τις επιδοτήσεις, πάντα οι ισοδομικές μεταφορές ήταν κάτι το οποίο σαν τα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε κανείς να το πειράξει. Για να δούμε τι θα γίνει στο Στασβούργο. Ελπίζω να καταφέρουμε μια αυθεντική ευρωπαϊκή αγορά γιατί έχουμε παρακαλοπιάσει τα κράτη-μέλη στο παρελθόν. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε στάση. Κύριε Στέριξ, ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο, ιδίω για αυτέ τι καθόλου ερετικές απόψεις που το στο τέλο. Τικάω, παρακαλώ ένα δίλεπτο. Η κυρία Τικάω. Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη σε αυτά τα δίλεπτα, στα ρουμανικά. Έχω δύο ερωτήσεις. Συγχαρητήρια, Υπουργέ, γιατί είσαστε ένας από τους πρόεδρους του Συμβουλίου που προσπαθείτε να ρυθμίσετε τα θέματα των εμπορευματικών μεταφορών, των μεταφορών για τις εσωτερικές πρωτές οδούς. Για πέστε μας τι πρόοδο, τι πρόοδος έχει ε, επιτευχθεί στο Συμβούλιο. Επίσης για πέστε μας όσον αφορά την οικονομική πολιτική αλλά και τις δημοσιομικές προοπτικές σε σχέση με την πολιτική των μεταφορών. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δημοσίευσε κατά την Προεδρία σας την ε, Λευκή Βίβλο, περιμένουμε, ούτε τις προοπτικές. Εδώ όμως τα έχουμε ήδη αυτά συζητήσει και το Συμβούλιο. Μάικλ, θέλεις να το λόγο ε, σαν, σαν αυτό που άκουσες. 30 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο χάνονται για, από το ΦΠΑ τον, και την, μάλλον, συγγνώμη, 30, δισεκατομμύρια ε, ε, δαπανώνται για την κυροζήνη και για το ΦΠΑ στις, ε, ε, στις αεροπορικές μεταφορές. Ε, αλλά οι θαλάσσιες μεταφορέ είναι φιλικέ προ το περιβάλλον. Μόνο εάν μπορέσουμε ε, να, έχουμε μια ενιαία φορολογία και αν μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα σκάφη και στι πλωτέ μεταφορέ, στου ποταμού. Okay. Ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Μάικλ. Υπουργέ, τώρα έχετε 10 λεπτά για αυτέ τι τόσο εύκολες ερωτησούλε. Εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο Υπουργό. Θα σας απαντήσω όσον αφορά τις παρατηρήσεις. Και ιδίω τα πιο αρνητικά από τα σχόλια τα οποία έγιναν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σας ξεκαθαρίσω το πώς έχει η κατάσταση να δούμε και για τους πόρους που έχουν δεσμευτεί όσον αφορά την Ευρωβινιέτα. Γιατί πρόκειται για κάποια πάρα πολύ δύσκολη επιλογή που να κάνουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια λύση συνεδρική Οι Υπουργοί Μεταφορών και αυτοί πιέζονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και άλλους και έχουν υποθεί εξής τάσεις. Πρώτον, υπάρχουν κάποιοι υπουργοί μεταφορών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ό,τι τυχόν είναι διαθέσιμο. Άλλοι πιστεύω να πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια φορολογική πολιτική και, και τα έσοδα αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία και να χρησιμοποιούνται για τις δημόσιες μεταφορές. Και πρέπει να τρίτη ομάδα υπουργών μεταφορών που ανησυχούν τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας τους και επομένως είπαν ότι όσα έσοδα προκύψουν από την Ευρωβινιέτα, αυτά θα πρέπει να διατεθούν για την εμπορική, για την πολιτική μεταφορών ε, στα κρατημέλη. Επομένω είχαμε τριπλή διάσπαση εν μέσω των Υπουργών. Δεν θέλουμε μαζί με τα ξένα και τα χλωρά, θέλουμε κάτι να βγει από αυτόν τον προβληματισμό. Πάντως δεν μπορώ τώρα να εμπιστεύω σε λεπτομέρειε. Νομίζω το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Και η Ευρωβουλευτή δεν θέλουμε να πέσει στο κενό σαν ιδέα. Τώρα, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με τον προπολισμό είχαμε πρόβλημα. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, δεν καταφέραμε πολλά. Και νομίζω ότι τελικά καταλήξαμε σε κάποια άτυπη συμφωνία που θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο. Όλα αυτά βεβαίως, επί Ουγγλικής Προεδρίας, με την οποία όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Τον Ιούνιο δεν θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε τα συμπεράσματα της Προεδρίας. Οπότε να υπάρχει κάποιος βαθμός βεβαιότητας ότι το περιεχόμενο της Λευκής Βίβλου που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θα εγκριθεί και θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις από αυτού για το πρώτο ήμιση του έτους. Τώρα, τι είπε ο κύριος Κράμερ, είπε για τις διαφορετικές επιλογές. Τις ε, επιλογές που είχε το Βέλγιο, ότι τελικά επέλεξε κυβέρνηση. Ε, επ' αυτό έχω να σας πω ότι η αφετηρία μας ήταν ότι η Ευρωβινιέτα δεν θα έπρεπε να αποτελεί έναν παραπάνω φόρο, ε, ένα παραπάνω γραφειοκρατικό εμπόδιο. Επ' αυτής της βάσης κινηθήκαμε. Και τώρα για τον κύριο Κράμερ πρέπει να σας πω, αλλά και για άλλους, ότι η πολιτική συγκυρία είναι τέτοια στο Βέλγιο που στην αρχή οι περιφερειακές κυβερνήσεις θέλαν να περάσουν κάποιο μέτρο για τις οδικές μεταφορές. Τελικά διαμορφώθηκαν τρεις διαφορετικές επιλογές ή βινιέτα αλλά ελετικά και άλλοι θέλανε να ε, ισχύει σαν κριτήριο ο αριθμός χιλιόμετρων που έχει ταξιδέψει το όχημα. Τελικά υπερέχει η λύση του υπολογισμού βάσει του αριθμού χιλιόμετρων που έχει ταξιδέψει το όχημα. Όσοι δε ήταν αυτές τη ιδέα, αυτής εξ αρχή αυτή είπαν ότι το κόστο θα αυξηθεί. Να ληφθεί υπόψη το πόσο έχει χρησιμοποιηθεί το όχημα, πόσο καθαρό είναι το όχημα, πόσο φιλικό στο περιβάλλον. Ήδη έχω συνοηθεί από αυτού με του υπουργού μεταφορών, του υπουργού κινητικότητα. Του εξήγησα τι έχει εγκριθεί ήδη και είπα ότι τώρα συζητείται στο Συμβούλιο κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οπότε Ελπίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος της Ουγγρικής Προεδρίας θα έχουμε μία σαφή ιδέα του πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. να αποφευθούν οι επιπλέον αχρίαστε δυσκολίε είπαμε, μεταξύ των περιφερειακών κυβερνήσεων και ευρωπαϊκού επίπεδου αποφάσεων, όλα θα πρέπει να είναι συμβατά με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην είναι συμβατότητα. Θα πρέπει να ισχύουμε το 2013. Κράμερ όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα ή την συμβατότητα μεταξύ οδικών και στερεοδρομικών μεταφορών. Αυτά τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Και συμφωνώ για το τι ισχύει για τους δρόμους και τα έχω συζητήσει με εκπροσώπους του κλάδου αλλά και με εκπροσώπους των οδικών μεταφορών, ο καθένας φυσικά μένει πιστό στις θέσεις του να λάβουμε υπόψη τι ισχύει τώρα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν είναι και τόσο αθέμητος, δεν είναι τόσο ιδιώδης κατάσταση όσον αφορά τον ε, ανταγωνισμό. Κάτι, τίποτα δεν είναι τέλειο σε αυτόν τον κόσμο και ε, επομένως δεν μπορούμε τη μια στην άλλη να πετύχουμε το τέλειο. Και το ξέρουμε. Τα έχουμε δε συζητήσει με τους εμπλεκόμενους και κάποιες βασικές αρχές θα πρέπει να ισχύουν σε όλου του είδους τις μεταφορές. Να έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση και δικαιότερο ανταγωνισμό. Υπάρχουν κάποια θέματα πάρα πολύ δύσκολα, όπως και τα θέματα της μόλυνσης και στις ελληνικές μεταφορές. Επομένως, εδώ θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά το αν θα πετύχουμε εναρμόνιση. Γιατί έχουμε το θέμα της Ευρωβινιέτας. Δύσκολα να πετύχουμε το... αυτό το οποίο θέλουμε. Δηλαδή, να είναι δίκαιες οι συνθήκες του ανταγωνισμού γιατί είναι γνωστό ποια είναι τα δυνατά σημεία σε κάθε είδος μεταφορών ε, αλλά δεν είναι πάντοτε σαφές που αγγείται τα πλεονεκτήματα. Ε, και αυτά θα πρέπει να τους τα λέμε. Φαντάμε. και η κυρία Τίκαου για ιστορικές πλούτες οδούς αλλά και τις ε, θαλάσσιες μεταφορές, εμείς επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο εξή. Σε ένα νέο στοιχείο στην ε, πολιτική μεταφορών. Ε, Της παράκτητες μεταφορές. Για το πώς θα μπορούσαμε να οργανώσουμε καλύτερα την εσωτερική αγορά, να την κάνουμε πιο φιλική στο περιβάλλον. Και έτσι θελασσιές μεταφορές και οι παράκτητες μεταφορές και αυτές να εμπλέκονται περισσότερο στην υπόθεση της μεταφοράς αγαθών μεταξύ των μελών. Άρα το, το μελετήσαμε το θέμα, λάβαμε υπόψη τι έχει πει το Κοινοβούλιο, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τι πρακτικέ μεταφορέ, θα πρέπει να οργανωθούν καλύτερα. Χρειαζόμαστε συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών επίσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να συνεργάζονται μαζί μας, να εγκρίνουν ό,τι κάνουμε. Μας είπε ο κ. Φαντάμε για το ατύχημα που συνέβη στο Ρήνο και τα συζητήσαμε αυτά με τους Ουγγρούς συναδέλφους. Είπαμε δε ότι το Βέλγιο θα συνεχίσει να ασχολείται με τα θέματα θαλασσιών μεταφορών. είναι πάρα πολύ σημαντικό ποτάμι, επομένω οι Ούγγροι δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα σοβαρά. Επομένω, ε, σίγουρα θα είναι θέμα οι μεταφορέ από τα ποτάμια. Τον Απρίλιο θα έχουμε μια τηλεσυνεδρία στη Βουδαπέστη. είναι τα θέματα που θα συζητηθούν τον Απρίλιο σε αυτή τη συνάντηση και αύριο θα έχετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες επί όλων αυτών. Για τον IMO Όχι, δεν λέω φαντά. Ούτε φαντάμε, θα Α, καλά. Καλά, ξέρετε ότι σε εσάς μιλάω πάντως. Εσάς εννοούσα. Όσον αφορά επομένω το 0,1% της μείωση του IMO, δεν ξέρω τι πας Και... και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Σαν συντελεστής. Αυτό θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό σε αυτές τις μεταφορές. Επομένως, είναι, είναι απότομη η μείωση. Θα έπρεπε πριν το 0,1 να κατέβουμε στο 0,5 και μετά να κατέβουμε κι άλλο. Πρόκειται για μια απόφαση της αρχής που θα έχει συνέπειες ε, πολλαπλές. Και το θέμα είναι το κόστος τώρα, πώς θα αυξηθεί. Έτσι θα πρέπει να το δει κανείς. Τι αντίκτυπος θα υπάρχει από πλευράς οικονομικής. Άλλο το τι θα γίνει πλευράς περιβάλλοντος και θα γίνει πλευράς οικονομικής. Κάποιες κυβερνήσεις θα έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν και πάρα πολύ η ευρωπαϊκή προσέγγιση, να δούμε όμω πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πριν να πρώτα, θα πω για τα εξωτερικά κόστη, που κάτι να αναφέρει και ο κύριο Στέρεξ. Μίλησα γι' αυτό. Όταν σας έλεγα για την Ευρωβινιέτα και για τα δεσμευόμενα κεφάλαια, το, το earmarking οι δύο υπουργοί οικονομικών πάντοτε θα έχουν λόγο. Ιδίω όπω είναι σήμερα η κατάσταση. Και όσον αφορά τα θέματα μεταφορών, δεν μπορέσαμε να σημειώσουμε όσο πρόοδο θέλαμε. Το ξέρουμε. Οπότε και την επομένη εβδομάδα ελπίζω ότι θα γίνει η αρχική ανταλλαγή απόψεων με τους Ούγγρους Συνάδελφου. Αυτά προ το παρόν. Με λίγα λόγια αυτά έχω να απαντήσω σε ερωτήσει που υποβάλλατε. Είχατε κάποια ερώτηση ή να απαντήσετε στον κύριο Κράμερ, συνάδελφε. Όχι, δεν είναι για τον κύριο Κράμερ. Ξέρει, ξέρει τι πρέσβευε ο κύριο Κράμερ. Όχι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό. Χωρί να είμαι σίγουρο για το πώ θα το κάνουμε. Γιατί έχουμε μετά του συντονιστέ, ξέρω εγώ. Αυτό, θα να πω στον κύριο Υπουργό, είναι πρώτα-πρώτα πάρα πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία για την συνάντηση κορυφή της Μπρίζ. Πολύ σημαντική. Και από ό,τι ξέρουμε υπάρχουν κάποια κρατημέλη που δεν προχωράνε όσο γρήγορα θα έπρεπε. Με το διοξίδιο και αυτά. Κύριε Υπουργέ, Έχετε τίποτα καινούριο μας πείτε όσον αφορά αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει στην αρχή της Προεδρίας, κάτι που το είπαμε και στην Κομισιόν. για τα θέματα τιμολογιακή πολιτική εταιρείων για του αεροδρόμου παντού στην Ευρώπη. Το είχαμε πει αυτό στην Κομισιόν. Μπα και θα μπορούσαν να πιέσουν τι εταιρείε τι αεροδρομικέ. Γιατί είναι δυνατόν κανεί με τον υπολογιστή να κλείσει εισιτήρια αεροπορικά και να πάει όπου θέλει στον κόσμο, αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε καν για την Ευρώπη στη, για τους ιδεοδρόμου. Αυτό αν το προωθούσε θα ήταν μεγάλη πρόοδο. Δεν έχετε να πείτε τίποτα βέβαια, ξέρω ότι καταρχήν μάλλον δεν γίνει απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Συγγνώμη που ακούστηκα λίγο κοινικός αλλά όταν οι εταιρείε, ε, οι μεταφορέ σιδηροδρομικέ ήταν στα χέρια του κράτου, υπήρχαν κάποιε ε, μεταφορέ οι οποίε ήταν πιο φθηνέ. Α πούμε, οι μεταφορέ φοιτητών. Τα φοιτητικά εισιτήρια ήταν πιο φθηνά για να μπορούν να πάνε ας πούμε, από το βορρά στο νότο τη Ευρώπη. Ένα εισιτήριο χρειαζόταν και μάλιστα σε μια πολύ καλή τιμή. Τώρα αυτές οι εταιρείε έχουν γίνει ανεξάρτητες και ανταγωνίζονται μια την άλλη, οπότε είναι αρκετά δύσκολο να λειτουργήσουν σε τόσο μεγάλο ε, πεδίο όπως είναι το ευρωπαϊκό και να δίνουν πιο φτηνά εισιτήρια. Βεβαίω αυτό το έχουμε υποβάλει στην Κομισιόν η Κομισιόν θα το κοιτάξει ε, περισσότερο για να δει αν μπορεί να γίνει κάτι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ κύριε Υπουργέ και εσάς και την, τους συνεργάτες σας κατά τη διάρκεια της, για την προεδρία σας. Όντως ήταν σημαντικό το πακέτο για τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, μερικές φορές μας δίνατε κάποια πράγματα, κάποιες φορές ε, ήταν λίγα και καλά αυτά που λαμβάναμε. Τέλος πάντων καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ξέρω ότι δουλέψατε πάρα πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της Προεδρία σα από του έξι μήνε. Σα ευχαριστώ που επανήλθατε σήμερα, που απαντήσατε στις ερωτήσεις, που ε, μας αναφέρατε τι έγινε στην Προεδρία σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Okay, uh, Ωραία. Συνάδελφοι, ως συνήθως, τέτοια εποχή, λέμε αντίο στον έναν υπουργό και λέμε καλώς ήρθες στον άλλον υπουργό. Επόμενο σημείο. Τουρισμός. Η κυρία Ιζαμπέλ Βάικμαν είναι η Υπουργός Τουρισμού. Να την καλωσορίσουμε. Okay, Ωραία, συνάδελφοι, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βάικμανς για να μας κάνει μια παρουσίαση των ε, πεπραγμένων της Βελγικής Προεδρίας στον τομέα του τουρισμού. Όποιος θέλει να συνεχίσει τη συζήτησή του, ευχαρίστως να το πράξει, αλλά εκτός της αίθουσας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε την Υπουργό. Έχετε το λόγο. Uh, okay, Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που είμαι και πάλι σήμερα εδώ. 198 ημέρες πέρασαν από τότε που ήμουν εδώ μαζί σας και παρουσίασα το πρόγραμμα της Προεδρίας μας ε, για τον τουρισμό. Αν θυμηθούμε έτσι λίγο πώς έγιναν τα πράγματα, είχαμε την στρατηγική ε, Λισαβόνας που άρχισε να τέθησε ισχύ. Ο, ε, ήταν σημαντικό ότι ο τουρισμός έγινε κομμάτι όλων των πολιτικών, ε, έτσι ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει και παραπάνω μέτρα πέρα από τους χειρισμούς που θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Βεβαίως όλα πάντα στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας. Στι εργασίες και σε ό,τι αφορά την, Βελική Βελική Προεδρία, εμεί ω. ένα από τα πρώτα, ήμασταν ένα από τα πρώτα κρατημέλη που δούλεψε σε αυτό το τρίο που λέμε ε, με τους Ούγκρους και τους Ισπανούς συναδέλφους και με τα αποτελέσματα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ο τρόπος αυτός, ο ανοιχτός τρόπος συντονισμού με τους ε, Ισπανούς, τους προκατόχους μας στην Προεδρία βοήθησε ώστε να υπάρξει μια δήλωση θα σας θυμίσω ότι έγινε αυτό στις 15 Απριλίου του 2010. Ε, η δήλωση αυτή έγινε, ως, ε, αποτέλεσε το μοντέλο για, τον, για την απόφαση που ελήφθη μετά για την πολιτική του τουρισμού στα πλαίσια πάντα της ε, πολιτικής επικουρικότητας. Η συντονιστική δράση λοιπόν της Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν μιλούμε για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, αν θέλουμε να τον βελτιώσουμε και αν θέλουμε να έχουμε μια, ε, ένα βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό και ένα βιώσιμο και υπεύθυνο μοντέλο τουρισμού. Τα κράτη-μέλη και σε αυτή την δήλωση πρότειναν ότι θα πρέπει να υπάρξουν νέα εργαλεία και για την πρόθεση του τουρισμού, αλλά και για τον τουρισμό και την πολιτική του τουρισμού θα πρέπει να ενσωματωθούν και τα υπάρχοντα εργαλεία που έχουμε για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Βεβαίως και η ανάπτυξη εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και πολύ σημαντικό επίσης και ένα από τα βασικά σημεία της Βελικής Προεδρίας ήταν ότι η ορατότητα της Ευρώπης θα πρέπει να βελτιωθεί επίσης. Το κείμενο αυτό τότε βοήθησε σε πολλές διαβουλεύσεις της Κομισιόν για, την, για να προετοιμαστεί η ανακοίνωση. Η Βελική Προεδρία ήδη από τον Ιούνιο είχε τη δυνατότητα να δει το, το σχέδιο αυτό της ανακοίνωσης και πολύ γρήγορα μπόρεσε να αξιολογήσει την όλη δυναμική που προέκυψε από την ανακοίνωση αυτή και από την Κομισιόν αλλά και τα κρατημέλη μπόρεσαν να ενεργοποιηθούν στον τομέα αυτό έτσι ώστε και η Κομισιόν στις 30 Ιουνίου του 2010 να μπορέσει να δημοσιεύσει την ανακοίνωση αυτή. Την ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας την αναφέρω, ε, η οποία αναφέρεται σε τέσσερις συγκεκριμένους άξονες. Ανταγωνιστικότητα, ποιότητα, βιωσιμός τουρισμός, ενσωμάτωση των ε, εργαλείων στον τομέα της πολιτικής, του τουρισμού και βεβαίως βελτίωση της εικόνας του τουρισμού στην ε, Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί ήταν οι τέσσερις ε, άξονε. Ε, η ανακοίνωση έπρεπε να είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβρη, αλλά έγινε στις ε, αρχές του, της Προεδρίας μας, πήγαμε γρήγορα, ε, οπότε μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Γιατί έτσι μπορέσαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα, πιο απτά μέτρα, να τα επεξεργαστούμε, να τα υποβάλουμε και αυτή τη ε, διαδικασία που είχε ξεκινήσει τότε, να την ξεκινήσουμε, να την ενισχύσουμε και να την προχωρήσουμε. Έτσι ώστε ό,τι υπήρχε μέχρι τότε να μπορέσει να αναχθεί και στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, πολιτική του ε, τουρισμού. Στις 30 ε, Ιουλίου ήμουνα εγώ εδώ και ήταν καλό που είδα ότι και από την πλευρά του Κοινοβουλίου υπήρχε, μεγάλη, υπήρχε πολύ μεγάλη αποδοχή και θετική άποψη για την κοινοποίηση αυτή της, για την ανακοίνωση της Κομισιόν. έτσι ώστε να δούμε ότι όντως ε, ήταν σωστή η προσέγγιση που είχαμε ακολουθήσει. Θέλαμε λοιπόν να έχουμε σύντομα αποτελέσματα τα οποία να μπορέσουν να συμφωνηθούν και αυτό σας είχα πει εγώ εδώ στις 13 ε, του Ιουνίου μετά είχαμε τον, ε, τις ε, καλοκαιρινές διακοπές και τον ε, Σεπτέμβρη που επανήλθαμε όλοι, εργαστήκαμε γρήγορα έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε τα περισσότερα κρατημέλη σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος μετά τον επεξεργαστήκαμε και υπευλήθη από τη δική μας μεριά και μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και μάλιστα περήφανοι θα μπορούσα να πω γιατί έχουμε, είχαμε το πρώτο επίσημο Συμβούλιο Υπουργών κατά τη διάρκεια της, προ, της μας, Υπουργών Τουρισμού και για πρώτη φορά ε, καταλήξαμε σε μια επίσημη απόφαση. Αυτό έγινε στις 12 Οκτωβρίου του 2010. Έγινε στο Λουξεμβούργο ε, η υπουργική αυτή διάσκεψη και όχι εδώ στις Βρυξέλλες. Υπήρξαν λοιπόν αυτά τα ε, συμπεράσματα, συμφωνήθηκαν, εγκρίθηκαν στα πλαίσια και τα οποία έθεσαν το πολιτικό πλαίσιο για τη, για τη μελλοντική πολιτική τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε περίπου, είχαν περίπου προταθεί 21 μέτρα. Τα, για τα κράτη-μέλη ήταν σημαντικό να είναι πιο συγκεκριμένα τα μέτρα αυτά, αλλά έπρεπε να υπάρξει και μία κατηγοριοποίηση, μία θέση προτεραιοτήτων. Για να δούμε δηλαδή ποια θα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν πρώτα και ποια θα είναι τα μέτρα που δεν επήγουν τόσο πολύ. Και επίσης έπρεπε να δούμε πολύ συγκεκριμένα με ποιον τρόπο θα, επί, θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα αυτή η πρώτη πρόταση, αυτό το πρώτο σχέδιο πήγε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού το, στη Μάλτα το Νοέμβρη, παρουσιάστηκε εκεί και έγινε η πρώτη διαβούλευση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ε, δόθηκε η εντολή να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση, πρώτη έκθεση αξιολόγησης το 2013 για να δούμε τελικά πού έχει φτάσει η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και πόσο έχει προχωρήσει. Υπήρχαν και άλλα σημεία σημαντικά στα, στα συμπεράσματα. Η ποιότητα, ας πούμε, ο βιώσιμος τουρισμός, ε, ο πολιτισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός που επίσης είναι σημαντικός, η καινοτομία, τεχνολογική δηλαδή, τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και ολοκλήρωση, ενσωμάτωση των χρηματοδοτικών μέσων τα οποία βεβαίω άπτονται περισσότερο ε, της πολιτικής, ε, στην πολιτική πτυχή της, του τουρισμού. Επίσης η εικόνα και η ορατότητα της Ευρώπης, η εικόνα της Ευρώπης προς τα έξω. Μπορέσαμε να ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό και με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού αλλά και με τη δημιουργία του προγράμματος που υπήρξε και που ασχολήθηκε αποκλειστικά με το θέμα αυτό. Βεβαίως ήταν ε, ο στόχος μας ε, ο υπεύθυνο και ποιοτικό αλλά και βιώσιμος τουρισμός. Εδώ μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε αυτή την αρχή στα συμπεράσματα. Ήταν ένα σημαντικό λοιπόν τμήμα αυτό των συζητήσεων του φόρουμ και η Βελγική Προεδρία ήταν πολύ ικανοποιημένη που μπόρεσε να ε, επηρεάσει και, και κατάλαβε ότι και η Κομισιόν μπόρεσε να υπογράψει την ε, συγκεκριμένη ε, απόφαση, η οποία ήταν πολύ σημαντική για να τεθούν τα κριτήρια για τον βιώσιμο τουρισμό. Ε, πολιτισμός και τουρισμός, επίσης σημαντικό θέμα. Και εδώ μπήκε, και το θέμα αυτό μπήκε στα συμπεράσματα. Συζητήσαμε και για τον πολιτισμό γενικώ και για το πώς αυτός μπορεί να συνδεθεί με τον τουρισμό. Ε, μπόρεσαμε λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να δούμε την προσθέμενη αξία που μπορεί να προκύψει από τον πολιτιστικό αυτό τουρισμό και να μπορέσουμε να τον υποστηρίξουμε. Επίσης, ανταλλαγή. Η ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών, Πρέπει να δούμε ποια είναι η διαδικασία, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα, είναι η, ποια είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τουρισμό και αυτό συζητήθηκε στο φόρουμ. Επίσης, Είχαμε πάνω από 400 συμμετέχοντες στο φόρουμ. Έγινε και άλλη μία συνάντηση εργασία μεταξύ κρατών μελών. Πάνω από 17 κρατημέλη έλαβαν μέρος. Και αυτό τονίζει ακόμη περισσότερο τη σημασία του τουρισμού για όλα τα κρατημέλη και για το, για το ευρωπαϊκό επίπεδο βέβαια. Για πρώτη φορά μπορέσαμε να έχουμε και μία γνωμοδότηση για, το πρώτο, για την πρώτη φάση της εφαρμογής, την οποία επέβαλε η Κομισιόν. Στις 3 Δεκεμβρίου η Κομισιόν ε, μέσω της γραπτής διαδικασίας ζήτησε, τις, παρατηρήσεις από τα κρατη για, αυτή, για αυτό το πρώτο πρόγραμμα. Ήταν σημαντικό λοιπόν να έχουμε απαντήσεις από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να έχουν αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οπότε υποθέτω ότι θα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία αξιολόγηση του από την Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν ότι έγινε αρκετά καλή και απρόσκοπτη εργασία ε, και στα πλαίσια τη ε, Βελγική Προεδρία. Νομίζω ότι παραδώσαμε απρόσκοπτα και τη Κιτάλη στην Ουγγρική Προεδρία, η οποία επίση θα λάβει υπόψη τη όλε αυτέ τι παρατηρήσει έτσι ώστε να μπορέσει και να τις βελτιώσει και να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους ε, μήνες και χρόνια και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερως ευτυχείς που δημιουργήσαμε τη βάση, θέσαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο τώρα η πολιτική ευρωπαϊκού, ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού μπορεί να ε, εφαρμοστεί, μπορεί να βελτιωθεί. Βρήκαμε συμβιβασμού ε, μέσα στα 27 κράτη-μέλη, μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάποια από τα συμπεράσματα και τώρα έχουμε αυτή τη βάση και τη δυναμική την οποία μπορεί να προωθήσει η Ουγγρική Προεδρία. Επίσης, χαιρόμαστε για τις, ε, και προσβλέπουμε στις περαιτέρω εξελίξεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε την στήριξή μας και, στου, και στους Ούγγρους συναδέλφους αλλά και στην ε, Τρόικα των ε, Προεδριών. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο χρόνο, Πρόεδρε. Αυτά σύντομα από μένα για το τι έγινε τους τελευταίους μήνες. Ευχαριστώ.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 Okay. Καλώς. Τρία λεπτά. Πρώτος, Φιντάντζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό για τους έξι μήνες της δουλειάς της. Δεν ήταν τόσο εύκολο να οικειοποιηθεί κανείς ένα τέτοιο θέμα, ένα νέο θέμα το οποίο, είναι κυρίως, το οποίο προηγουμένως ε, εντασσόταν στην επικουρικότητα. Οι νέες αρμοδιότητες που ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας για τον τουρισμό μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέμβουμε με θετικές δράσεις, συντονισμό και ανταλλαγή θετικών πρακτικών. Μας περιορίζουν όμως ως προς την ομοθετική δράση, διότι όπως γνωρίζετε δεν προβλέπεται η δυνατότητα δράση σε νομοθετικό επίπεδο. Τώρα, το ότι δόθηκε μια όθηση και εντάχθηκε ως προτεραιότητα στους στόχους της Βελγικής Προεδρίας και ο τουρισμός ήταν πάρα πολύ θετικό πράγμα. Και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας ήταν και το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική δήλωση και το φόρουμ της Μάλτας μετά. Πολύ σημαντική ε, ε, συνάντηση μαζί με τους ε, tour operator και τα κράτη-μέλη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος ε, θεωρού, προχώρησαν σε ανακοινώσεις με πάρα πολύ φιλόδοξα σχέδια. Όλοι έχουμε αναλάβει, εγώ ως εισηγητή, όλοι οι εισηγητές, έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτή τη νέα στρατηγική για τον τουρισμό. Εμείς έχουμε βέβαια εδώ κάτι το απαγοητευτικό είναι το θέμα των κονδυλίων, δεν έχουμε λεφτά. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή των θετικών πρακτικών, αλλά πρέπει όμως να παλέψουμε στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές μέχρι το 2013 να έχουμε ειδικέ γραμμές για τις πολιτικές τουρισμού, διότι αλλιώς δύσκολα μπορούμε εμείς να, συμπληρώ, να ολοκληρώσουμε αυτές τις 21 δράσεις που έχει προβλέψει η Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε ειδικέ γραμμές στον προϋπολογισμό διότι αλλιώς οι 21 δράσεις που πρόβλεψε η Κομισιόν αλλά και άλλες προτεραιότητες που μπορεί να προκύψουν από το Κοινοβούλιο θα μείνουν ανέφικτες. Ο Υπουργός και η Ουγγρική Προεδρία θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους μαζί με την Κομισιόν ούτως ώστε να δώσουν και τα απαραίτητα κονδύλια διότι έχουμε ελάχιστα κονδύλια για τον τουρισμό. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν μια μεγαλύτερη ορατότητα σε όλους αυτούς τους πόρους ε, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι στα διάφορα ταμεία, στα, στα διάφορα διαρθρωτικά ταμεία, στο κοινωνικό ταμείο κλπ. Πρέπει αυτά τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν για την τουριστική ανάπτυξη. Πέρα όμως από αυτά τα κονδύλια, τα οποία αφορούν στον τουρισμό αλλά δίνονται από τα ταμεία, πρέπει να έχουμε και δικές μας αυτόνομες γραμμές στον προπολογισμό. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα βοηθήσει να καταλήξουμε σε αυτόν τον στόχο. Τελειώνω τώρα πρόεδρε, τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσουμε την έκθεση και θα ήθελα να τονίσω εδώ δύο προτεραιότητες που αποτελούν αρχή και το τόνισε και η υπουργό. Πρώτον, κατάρτιση. Πρέπει να επενδύσουμε πολύ στην κατάρτιση. Όχι μόνο στις παραδοσιακές, ε, ε, παραδοσιακές ε, δραστηριότητες, αλλά σε νέες δυναμικές που θα δώσουν μεγαλύτερη ορατότητα στον τουρισμό. Επίσης, τεχνολογική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε εμείς να παραμείνουμε στο παραδοσιακό μοντέλο τουριστικής επιχείρησης. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάτι το σύγχρονο, το μοντέρνο. Ο κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Βελγική Προεδρία ευτύχησε να εγγράψει στον απολογισμό δράστης για τα θέματα του τουρισμού την πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Τουρισμό, καθώς επίσης και την σε εξέλιξη ευρισκόμενη συζήτηση για τη σύνταξη της πρώτης έκθεσης του Κοινοβουλίου μας για τον Ευρωπαϊκό Τουρισμό, μέσα στη νέα πραγματικότητα την μετά τη Λισαβόνα, όπου ε, έχουμε πλέον ως Ευρωπαϊκή Ένωση την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να στηρίζουμε, να συντονίζουμε και να συμπληρώνουμε τη δράση των κρατών μελών. Φοβάμαι ότι δεν ε, θυμόμαστε πάντοτε ότι ο, ο τουρισμός είναι μια ύψιστη της σημασίας τουριστική αλλά και κοινωνική δραστηριότητα για την Ευρώπη. Φοβάμαι ότι αγνοούμε ότι στον τουρισμό οφείλουμε το 10% περίπου του ακαθάριστου ευρωπαϊκού εισοδήματος, καθώς επίσης και τη διασφάλιση του 12% των θέσεων εργασίας. Αναφέρεται σε μια πολύ μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων, αλλά είναι παράλληλα και ο βασικότερος τρόπος προσέγγισης και αλληλοκατανόησης και γνωριμίας των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι πώς μεγιστοποιούμε, πώς εξειδικεύουμε ένα σύνολο συγκεκριμένων πολιτικών για την τουριστική μας ανάπτυξη, αλλά και πώς εξασφαλίζουμε συγκεκριμένες συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξουμε αυτές τις πολιτικές που δεν μπορούν παρά στόχο να έχουν την πρόθεση ενός άλλου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης ποιοτικά βελτιωμένου, βιώσιμου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Mr. Ugias for uh, ALD, please. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν ε, θα κάνω, δεν θα βγάλω λόγο. Ερωτήσεις θα απευθύνω για να πάρω και απαντήσεις. Κοιτάστε, έξι μήνες περνάνε πάρα πολύ γρήγορα όταν έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Αλλά θα ήθελα να ξέρω, στα πλαίσια του Συμβουλίου, Το θέμα του τουρισμού συλλογικά εξετάστηκε πρόσφατα από την Κομισιόν. Πιο συγκεκριμένα θα ρωτούσα στις συζητήσεις που γίνονται μέσα στο Συμβούλιο για το θέμα της χρηματοδότησης υπάρχει ένα σημείο ξεκινήματος Βασίζεστε κάπου ή πρέπει ακόμη να το διαμορφώσετε αυτό το σημείο. Δεύτερο, η ανακοίνωση ευθυγραμμίζεται με την Ευρώπη 2020 ή πρέπει να βελτιωθεί ακόμα. Τρίτη ερώτηση. Ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε εσείς ότι θα οριμάσουν το, κατά το επόμενο εξάμεινο. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο πήρατε εσείς, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα συνεχίζονται πλέον στο δεύτερο εξάμεινο και θα αναπτυχθούν. Ο κύριος Κρέμερ για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. η στρατηγική της ε, Λισαβόνας εφαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό γιατί βασίστηκε στον ε, τουρισμό ήδη. Ε, ξεκίνησε μάλλον από την, με την αρχή που κάνατε εσείς με τον τουρισμό. Ήδη λοιπόν αυτό είναι κάτι θετικό. Ακούσαμε όμως πολλά από όσα είχαμε ήδη ακούσει. Ακούσαμε πολλές φορές αυτό τη λέξη βιώσιμος, βιωσιμότητα. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά, αλλά μεταξύ πράξεων και δράσεων, ε, υπάρχει μεγα... Ε, μεταξύ δράσεων και λόγων, συγγνώμη, υπάρχει μεγάλη απόσταση μέχρι, από το καλά είναι τα λόγια, αλλά μέχρι να φτάσουμε στα έργα και στα αυτά προγράμματα, εκεί είναι, εκεί είναι τα δύσκολα. Γιατί ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι ο τουρισμός μπορεί να καταστρέψει τον τουρισμό. Όχι μόνο την γεωργία, αλλά και την οικονομική βάση και, χωρίς, και μόνο από τον τουρισμό δεν μπορεί κανείς να ζήσει. Ούτως ή άλλως αυτό είναι σαφές. Έχω ένα ερώτημα όμως. Ο τουρισμός έχει να κάνει με τις ε, μεταφορές. Και ξέρουμε ότι οι μεταφορέ επίση μπορούν να γίνουν με οικολογικό τρόπο. Για να γίνει όμω αυτή η σύνδεση, είτε μέσω της, ε, στους διάφορους ε, τουριστικούς προορισμούς, και ένα μπορεί να υπάρξει ένα ε, ένας κατάλογος που να λέει ότι αν ταξιδέψετε με αεροπλάνο ε, θα έχετε τόσο ε, ε αρθρακικό αποτύπωμα, αν έρθετε με τρένο θα έχετε τόσο. Ε, πώς θεωρείτε ότι μπορείτε, μπορεί να γίνει αυτό, αν μπορεί να γίνει εσείς. Και επίση, χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνε προ τη λαθασμένη κατεύθυνση. Οπότε δεν υπάρχει καμία α, βιωσιμότητα στον τουρισμό και μάλιστα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο το, η κλιματική κατάσταση που επικρατεί. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε και ποια είναι αυτά τα προγράμματα του τουρισμού που πάνε προ σωστή κατεύθυνση. Γιατί καλά να χρηματοδοτούμε, αλλά να χρηματοδοτούμε και τα σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την Υπουργό για όλα όσα έκανε. Ε, νομίζω ότι όντως με την με τις, με την συνθήκη της Λαβώνας μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα. Νομίζω ότι είναι, έχει υπάρξει πάρα πολύ καλός ε, τρόπος για να, τονίσει, να τονιστεί η σημασία της, ε, του τουρισμού, αλλά όταν μιλάτε για αύξηση αρμοδιοτήτων, όταν το Συμβούλιο συζητά για, την, ε, το συντονισμό, έχει υπάρξει κάποια αξιολόγηση της, της κρίσης, το πώς έχει επηρεάσει η κρίση των... Ε, τον, ε, τον τουρισμό, πώς αν έχουν μειωθεί ας πούμε οι ώρες ταξιδιού, πώς έχει ε, επιβαρύνει τους ίδιους τους επιβάτες η κρίση. Και επίσης πολλές φορές οι γειτονικές χώρες έχουν αντικρουόμενες πολιτικές η πολιτική ενός, του ενός κράτους μέλους μπορεί να επηρεάσει τον άλλον, είτε είναι ε, φορολογικό δίκαιο, είτε είναι οτιδήποτε. Έχουν γίνει καθόλου τέτοιες συζητήσεις στο Συμβούλιο. Έχετε δει αυτές τις προκλήσεις, ειδικά και για το 2011, για τον τουρισμό. Και άλλο ένα ερώτημα. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Κράμερ και, την, ε, και τις μεταφορές. Πέρσι, ως αποτέλεσμα του, της, ε, του ηφαιστείου, Βεβαίω, εσεί τότε δεν είχατε προεδρία, ε, προετοιμαζόσασταν όμω. Καταλήξαμε στο ότι το στο τέλος του έτους επηρεάστηκε πάρα πολύ ο, ο τουρισμός. Επίσης, όταν έφτασε το τέλος του έτους είχαμε πολλές χιονοπτώσεις και επίσης ε, επηρεάστηκε ο τουρισμός. Υπάρχει κάποιο, κάτι που μπορούμε να κάνουμε για το, δηλαδή με τις ασφαλιστικές εταιρείες υπάρχει κάποιο, κάτι που μπορούμε να κάνουμε ή απλώς θα επαφιέμεθα σε αυτές για την ε, ε, αντικαταβολή των ε, ζημιών που προκύπτουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσίασή της. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια, ήδη τα είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Είπατε ότι η εντολή αυτή περιείχε 21, 21 μέτρα. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι τομείς που ε, πλήττονται από αυτά τα μέτρα. Ε, μας είπατε τέσσερις, αλλά μας είπατε για 21 μέτρα και θα θέλαμε λίγες περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, οι, χρηματο... οι γραμμές χρηματοδότησης. Η Λισαβόνα είναι αυτή που είναι, η συνθήκη είναι αυτή που είναι τώρα και ο Ιταλός συνάδελφος που πήρε πρώτος το λόγο το είπε. Δεν έχει να κάνει άμεσα με την νομοθεσία αυτό, αλλά εάν μιλούμε για γραμμές χρηματοδότησης, τα κρατη δεν έχουν χρήματα. Από πού θα προέρχονται λοιπόν τα χρήματα αυτά για τις γραμμές χρηματοδότησης. Και χωρίς να θέλω να είμαι ιδιαίτερο κοινική, αλλά ο τουριστικός τομέας είναι ιδιαίτερος ανταγωνιστικός και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Όλα τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν το ένα το άλλο για να έχουν περισσότερους τουρίστες. Ίσως να πρέπει να υπάρξουν κάποια κριτήρια ε, το, βάσει των οποίων να πρέπει να ε, εξοπλίζονται ας πούμε τα ξενοδοχεία. Να ξέρεις δηλαδή ότι αν πας σε ένα ξενοδοχείο στην τάδε χώρα ή στην τάδε χώρα θα είναι η ίδια ποιότητα. Και πώς ακριβώς θα δουλέψει όλο αυτό το σύστημα. Δεν μιλώ για την συνεργασία. Όλοι ε, θέλουν να έχουμε καλή συνεργασία, συνεργασία κτλ. Αλλά όταν αρχίζουμε να μιλούμε για χρηματοδοτικά εργαλεία και χρήματα και γενικώ θέματα οικονομικά, ε, εσείς πώς ακριβώς βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Προς τα πού θέλετε, θα θέλατε να πάει όλο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι και κυβερνήσεις που δεν είναι στην ε, μεταβατική φάση μπορούν επίσης να ε, συνεργαστώ. Μιλώ για, τον, ε, για την Novum Tourismus μια ένωση γερμανόφωνων. Σας, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω γιατί κάνατε καλή δουλειά και δεν είναι εύκολο ο τομέα που αναλάβατε και από την αρχή και το πώς παρακολουθήσατε το θέμα. Ε, εντάξει, δεν ήταν και πολύ ε, περιορισμένα τα μέσα που είχατε στα διάθεσή σας, ήταν όμως ε, λίγα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολλά, τα καταφέρατε όμω. Το θέμα του χρηματο... ήταν πολύ ε, σημαντικό. Το είχαμε συζητήσει και με, το θέμα, και με τον τομέα των ε, μεταφορών αυτό και πώς θα γίνει η χρηματοδότηση. Υπάρχει κάποια σύνδεση μεγαλύτερη με, την, ε, με, το, ε, με τα διαθετικά ταμεία για την διασυνοριακή συνεργασία. Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια γραμμή ειδική μόνο για τον τουρισμό. Γιατί και στον, στον τουρισμό η παιδεία παίζει πολύ υποτιμημένο ρόλο, παρόλο που είναι σημαντική. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το τονίσουμε ακόμη περισσότερο. Εγώ έρχομαι από μια περιφέρεια που δεν θέλω καθόλου να καταστρέψουμε τη φύση, όπως λέει ο συνάδελφος Κράμερ. φυσικά και δεν πρέπει ε, στο όνομα του τουρισμού να τα εξυγχρονίσουμε όλα και να τα καταστρέψουμε όλα, αλλά το ερώτημα παραμένει. Εσείς στο μέλλον, σε σχέση με αυτό, όχι μόνο για τη βιωσιμότητα του τουρισμού, αλλά γενικώ για τον τομέα του τουρισμού, ε, μπορείτε να αγγιηθείτε με κάποιο τρόπο ότι θα υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, αλλά και σε ό,τι αφορά το δικαίωμα που έχουν να ενημερώνονται οι πολίτε. Γι' αυτό επανέρχομαι στο ερώτημα. Στο μέλλον, πώ βλέπετε εσύ την κατα... εσείς την κατάσταση να, εξελίσετε. να Μπορούμε να μιλήσουμε μία ενιαία φωνή για να μπορέσουμε να συνονιθούμε όλοι μεταξύ μας και να, έχουμε και, να κατανοούν οι πολίτες τι συμβαίνει αλλά και να μπορούν οι πολίτες να παρουσιάσουν καλύτερα την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Πολύ θετικό ε, είναι το γεγονός ότι είσαστε υπουργό τουρισμού. Κάποιες χώρες δεν έχουν καν υπουργό τουρισμού. Χαίρομαι λοιπόν που ήρθατε εδώ σήμερα και μπορούμε να συζητήσουμε. Έχω κάποια ερωτήματα για τη δική σας ε, εντύπωση, για το πώς θα, εξηγηθεί, πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Είπαμε για την ε, εικόνα και για την ορατότητα της Ευρώπης ό,τι αφορά τον, τον τουρισμό, αλλά μιλούμε για μια τεράστια ευρωπαϊκή αγορά τουριστών. Βεβαίω πρέπει να δούμε και εσωτερικά πώ μπορούμε να κάνουμε τα κρατημέλη πιο, πιο ελκυστικά, ελκυστικά, αλλά επίση πρέπει να δούμε και πώ θα γίνει και η Ευρώπη στο σύνολό τη πιο ε, ελκυστική. Ε, εντάξει, δεν έχουμε μόνο να προσφέρουμε την Ακρόπολη και τον πύργο της Πίζας. Ε, εντάξει, την πύλη του Βραδεμβούργου δεν την ανέφερα. Αλλά εσείς πώς ακριβώς ε, το σκέφτεστε, πώς μπορούμε δηλαδή να τονίσουμε και, άλλα, και άλλους τομείς, άλλους κλάδους ε, του τουρισμού, ας πούμε, ε, τουρισμό για συγκεκριμένες, για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, πολιτιστική κληρονομιά, για σπα, για ε, για κούρα ή για ε, για πράγματα που προς το παρόν στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερος ε, προβεβλημένα. Και τέλος, τουρισμός στις, σε προστατευόμενες περιοχές, σε προστατευόμενες ζώνες. όπου να μπορεί κανείς να φτάσει και, να, και παράλληλα βεβαίως να μην καταστρέψει αυτή την προστατευόμενη ζώνη, να έχει όμως και το δικαίωμα να κινηθεί μέσα σε αυτή. Ευχαριστώ. We need... Thank you. Thank you. I just... Ναι, θα το πω εγώ, αυτό που αφορά τους δρόμους, αλλά πρώτα δώσουμε το λόγο στην Υπουργό. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω Ελπίζω να μπορέσω να καλύψω τα ερωτήματά σας. Το θέμα των χρηματοδοτικών μέσων ήταν ένα από τα βασικά θέματα που ανέφεραν πολλοί από εσά. Ένα ερώτημα τέθηκε για το από πού, ποιο είναι το σημείο κίνησης και ποια είναι η ατμόσφαιρα που υπάρχει γενικώ στο Συμβούλιο και πώς το βλέπουν τα κράτη-μέλη, πώς μπορούν δηλαδή να ε, κινητοποιηθούν και, να, και συντονισμένα και συμπληρώνοντας το ένα το άλλο να προχωρήσουν. Είπα ότι έχουμε επιτύχει μεταξύ των 27 κρατών μελών έναν συμβιβασμό σε διαφορά τα συμπεράσματα τα οποία βασίζονται σε αυτή την κοινοποίηση την ανακοίνωση της Κομισιόν. Ε, Γενικώ πώς υπάρχει ένα πλαίσιο, ο συμβασμός προφανώς δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί, για να απαντήσω ε, συγκεκριμένα, γιατί φυσικά οι απόψεις των κρατών μελών είναι διαφορετικές, και εξακολουθούν να είναι διαφορετικές, ειδικά ας για τον ε, ρόλο της Ευρώπης στον τομέα του τουρισμού. Οπότε γι' αυτό ήταν ακόμη πιο σημαντικό να έχουμε ένα κείμενο, αυτά δηλαδή τα συμπεράσματα που τα έχουμε τώρα, τα οποία να τη βάση συμφωνίας συνεννόησης μεταξύ κρατών μελών. Μπορέσαμε λοιπόν να συμφωνήσουμε επί αυτών των συμπερασμάτων, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια μεθοδολογία, ένα πλαίσιο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, απόψεων, εμπειριών, έτσι ώστε να μπορέσουμε πάνω σε αυτά να προχωρήσουμε, να εξελιχθούμε και η, ε, βιώσιμη, πούμε, η βιωσιμότητα του τουρισμού να μπορεί να προκύψει ε, παντού, όχι μόνο όπου, υπάρχουν, ε, όπου υπάρχει ήδη, δηλαδή υπάρχουν κράτη-μέλη, περιφέρειες, οι οποίες ήδη ε, έχουν μια, πιο βιο, μια προσέγγιση πιο βιώσιμου τουρισμού, αλλά να μπορούμε αυτό να το μεταφέρουμε και αλλού. Να έχουμε δηλαδή υποδείγματα, καλές πρακτικές, παραδείγματα που να μπορούμε να τα ε, επιδείξουμε. Και έχουμε και την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού να έχουμε κριτήρια τα οποία να εφαρμόζονται χωρίς κατά ανάγκη να πρέπει να εμπλέκονται, να εμπίπτουν σε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Και είπα ότι υπάρχει και αυτή η συμφωνία μεταξύ Κομισιόν και Νέξτορ και ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνεται εκεί, α, μεταξύ αυτών των 21, είναι και ο κατάλογος αυτός με τα κριτήρια δηλαδή τι χρειάζεται για να υπάρξει βιώσιμος τουρισμός και πώς μπορούμε να κάνουμε την δική μας προπαγάνδα και εμείς υπέρ αυτού. Τώρα, ποια είναι αυτά τα 21 μέτρα, με ρωτήσατε. Είναι τα μέτρα που υπάρχουν στην ανακοίνωση. Είναι... Υπάρχουν οι τέσσερις άξονες που σας ανέφερα αυτοί οι τέσσερις βασικοί, βασικοί άξονες και για μας ήταν σημαντικό να τεθούν συγκεκριμένα, ε, να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι πυρήνες. Το ξεκίνησε αυτό η Κομισιόν, έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει από το 2011 και μετά και τώρα βεβαίως κατά τη διάρκεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας γιατί υπάρχει και αυτό το πρώτο σχέδιο εφαρμογής, το οποίο πρώτο, πρώτη φορά υπάρχει και είναι εντάξει και συμπεριλαμβάνονται όλα όσα τα κράτη-μέλη ζήτησαν και όλα όσα ζήτησαν οι ε, μπλεκόμενοι φορείς, όλοι οι stakeholders. Αυτό λοιπόν είναι ένα σχέδιο εφαρμογής, το οποίο προτάθηκε από την Κομισιόν και επί του οποίου μπορούμε όλοι να βασιστούμε και επί του οποίου όλοι συμφωνήσαμε. Οπότε θα δούμε πώς θα έχουν τα πράγματα μέχρι το 2013. Μπορούμε ήδη από τώρα να το δούμε εφόσον όλα αυτά που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό εφαρμοστούν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ε, εργαζόμαστε, το πλαίσιο αυτό που δημιουργήσαμε, το πλαίσιο των συμπερασμάτων. Ε, όλα τα κρατημέλη το στηρίζουν και ξέρουν ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να γίνει ό,τι γίνει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια των συμπερασμάτων θα πρέπει να προταθούν μέτρα από την Κομισιόν. Και έτσι θα πάμε βήμα-βήμα για να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε σε μια επιτυχή πολιτική τουρισμού, η οποία φυσικά θα την χάνει μόνιμου συντονισμού. Αυτό είναι σαφές. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδικασίας και ε, τη νιώθουμε αυτή τη δυναμική που υπάρχει. Βλέπουμε την, ε, ότι πρέπει να ενισχυθεί και η ε, ευαισθητοποίηση των πολιτών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί υπάρχει και οικονομική πτυχή, υπάρχει και κοινωνική πτυχή στον τουρισμό και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο αυτό γιατί όντω η πολιτική τουρισμού μπορεί και πρέπει να παίξει έναν ε, σημαντικό ρόλο, γιατί εμπλέκεται και στην ε, πολιτική για το 2020. Αυτό συζητήθηκε λοιπόν στο Συμβούλιο Υπουργών. Οι στόχοι είναι οι ίδιοι, δηλαδή η βελτίωση των προτύπων που αφορούν τον τουρισμό, ε, χρηματοδοτική ενίσχυση, ένας τομέας είναι ο τουρισμός όπου υπάρχει μεγάλη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι στόχοι που ούτως ή άλλως ε, περιλαμβάνονται και στη στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουρισμός και μεταφορές. Τι γίνεται και πώς υπάρχει, ποια είναι η διασύνδεση που υπάρχει. Φυσικά υπάρχει μεγάλη διασύνδεση. Πώς το διαχειριστήκαμε εμείς. Αυτό το θέμα το συνδέσαμε με τα συμπεράσματα λέγοντας ότι υπάρχει το κοινοτικό κεκτημένο το οποίο επίσης επηρεάζει πολύ τα πράγματα για το πώς θα εδρεωθεί μια πολιτική για τον, για τον τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς πολιτικής που επηρεάζονται από αυτό ε, πολιτική περιβάλλοντος, μεταφορών, ε, καταναλωτών, πολλά, πολλοί τομείς, οι οποίοι ήδη έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία σήμερα από ό,τι είχαν παλαιότερα. Και σε, αυτό το τομέα, και σε αυτή την κατηγορία είναι και ο τουρισμός. Και αυτό θα γίνει μέσω ε, κανονισμών, οδηγιών που θα φορούν τον τομέα του τουρισμού Και βεβαίω θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μα το τι θα σημαίνει για τον ευρωπαϊκό τουρισμό αν λάβουμε αυτό το μέτρο ή αν λάβουμε το άλλο μέτρο. Αυτά έχουν συμπεριληφθεί λοιπόν στα συμπεράσματα. Και εδώ η Κομισιόν κάνει την αξιολόγησή της, ε, κάνει λοιπόν έτσι μια, ένα σκάνινγκ όλων των στοιχείων για να, δουν, για να δει τι ακριβώς επηρεάζει την πολιτική τουρισμού, τι ακριβώς επηρεάζει τον, ευρωπαϊκό τουρισμό και πώς πρέπει τα πράγματα να προσαρμοστούν ή πώς πρέπει να, αλλαγού, να αλλάχθουν ή πώς πρέπει να προχωρήσουν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως συνδέεται και με την πολιτική για τις μεταφορές. Η, αναφέρεται την κρίση με το ηφαίστειο. Ε, στην ίδια κατηγορία ε, εμπίπτει και αυτό. πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση. Διαχείριση κρίσεων, έτσι όπως ήταν εκείνη με το ηφαίστειο. Γιατί αυτό έχει μεγάλη επίδραση στον τουρισμό. Φυσικά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Και βεβαίω όλα αυτά ε, συμπεριλήφθησαν και στη συζήτηση που έγινε με την Κομισιόν. Τώρα πάω στα θέματα της, ε, της Αυτό το θέμα της ενιαίας ποιότητας, το είπε και ο κ. Γκρός, το είπαν και άλλοι, όντως είναι σημαντικό, πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Υπάρχουν προτάσεις, οι οποίες ε, αναφέρθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού και νομίζω ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει λοιπόν μία βάση για να καθοριστούν κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε και να συμφωνήσουμε επί των κρατερίων αυτών. Δηλαδή η ε, ε, ε, τα ποιότητας για την Ευρώπη. Τώρα θα δούμε βέβαια, γιατί υπάρχουν πολλοί νομοθέτε εδώ στα διάφορα επίπεδα, περιφέρειες, Ευρώπη κτλ. Θα, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αλλά εδώ πρέπει να επεξεργαστούμε και να καταλήξουμε σε κάτι, το οποίο βεβαίω θα είναι σε θελούσια βάση πάντα. Και θα πρέπει να υπάρχει και ένα, ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Και αυτό ετέθη προς Στην ε, Γερμανία, στην Ελβετία, στη Γαλλία υπάρχει τέτοιο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Και στην Ισπανία επίσης, γιατί υπάρχουν και μεγάλοι πάροχοι ε, τουριστικών πακέτων κτλ. Αυτή λοιπόν η ετικέτα ποιότητας όσο θα μπορούσε να εισαχθεί ως ε, ένα βασικό στοιχείο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Η Ευρώπη έχει πολλά να προσφέρει, είπατε κι εσείς, ε, από πολιτιστικέ κληρονομιέ μέχρι οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα πρέπει όντω να δούμε και άλλε πτυχέ. Φυσικά θέλουμε βιώσιμο τουρισμό, θέλουμε ποιοτικό τουρισμό και θέλουμε να προωθήσουμε αυτό που έχουμε να προσφέρουμε. Και βεβαίω ο πολιτιστικό τουρισμό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτά νομίζω είναι τα τρία βασικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται ως βάση στα συμπεράσματα. Τώρα πάω στα χρηματοδοτικά, που είναι σημαντικά και για το Κοινοβούλιο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το έχουμε συζητήσει και στη ε, συζήτηση που έγινε για τα συμπεράσματα. Ε, κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας ήταν σαφές ότι δεν, ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε γραμμή για τον τουρισμό ως το 2013 από εκείνες τις προοπτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας ε, μιλά για συγκεκριμένη πολιτική τουρισμού. Βεβαίως ε, υπάρχει ακόμα μια, ένας δισταγμός από πολλούς ναι, αλλά αν κάνουμε κάτι καινούριο, σημαίνει καινούριο, καινούριες δαπάνες και έχουμε λίγα χρήματα και δεν φτάνουν τα χρήματα. Αυτό συζητούμε συχνά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά έγινε η συζήτηση και ο συμβασμός τον οποίο καταλήξαμε ήταν σαφής. Πρέπει, πρέπει να κινητοποιηθούμε και πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για τον τομέα του τουρισμού. Χωρίς χρήματα κανείς δεν μπορεί να κάνει καμία είδους, κανένας είδους πολιτική. Αυτό ισχύει και για τον ε, τομέα του τουρισμού. Είπαμε λοιπόν, ναι, θα υπάρξουν χρήματα ή θα πρέπει να υπάρξουν χρήματα για τον τομέα του τουρισμού και σε ένα δεύτερο επίπεδο είπαμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε πάλι κάτι από την αρχή, από το μηδέν, αλλά θέλουμε να υπάρξουν συγκεκριμένοι τομής στα πλαίσια των υπάρχοντων ε, ε, προοπτικών, των υπαρχουσών γραμμών για τον προπολογισμό, έτσι ώστε να επιλέξουμε τη σωστή κατεύθυνση και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για τον τουρισμό. Να εμπλέξουμε και τα διαρθρωτικά ταμεία, να εμπλέξουμε και το κοινωνικό ταμείο. Γιατί μπορούν, μπορεί να υπάρξει γραμμή για τον τουρισμό μέσα σε αυτά τα υπάρχοντα ε, χρηματοδοτικά μέσα. έτσι ώστε να μπορέσουν και οι Ευρωπαϊκοί Ένωση στο αλλά και οι περιφέρειες που ε, ε, υποφελούνται από το Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια. Είναι σημαντικό λοιπόν, έτσι ώστε να έχουμε και μια συνέχεια, μια συνέπεια ε, στον, σε ό,τι αφορά τους στόχους που θέτουμε και για τον τουρισμό και για το διαρθωτικά ταμεία και για το κοινωνικό ταμείο. Να έχουμε λοιπόν μια συνέχεια έτσι ώστε να επιτύχουμε το ότι ο τουρισμός θα δημιουργήσει νέα ανάπτυξη ε, να λάβουμε υπόψη μας και την οικολογική πτυχή και το περιβάλλον. Αυτά φυσικά δεν τα ξεχνούμε. Είναι βασικές αρχές οι οποίες ούτως ή άλλως προωθούνται και μέσω των ταμείων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα μπορέσει να είναι ένα ακόμα ε, πλέον έκτημα για τη μελλοντική πολιτική για τον τουρισμό. Αυτή είναι η αρχή που συμφωνήθηκε από τα 27 κρατημέλη. Αυτή ήταν, ε, αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης εφόσον θέλουμε να μιλούμε συγκεκριμένα για τα, ε, για τα κονδύλια. Η αρχή λοιπόν νομίζω ότι είναι σχετικά σαφής. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι ε, απήντησα σε όλα. Αν όχι, αν ξέχασα κάτι, θυμήστε το μου και ευχαρίστως να σας απαντήσω. No. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και όπως είπα και στον συνάδελφό σας, σας ευχαριστούμε εσά και το επιτελείο σας για όλες τι προσπάθειε του τελευταίου εξαμήνου τη Υπηρετικής Προεδρία Ε, <clears throat> τα πάντα και στο μέλλον, ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και πάλι ευχαριστούμε. Okay, colleagues. Okay, colleagues, the next... Πολύ ωραία, συνάδελφοι. Το επόμενο θέμα της διάταξης τώρα είναι το κείμενο για την πολιτική συνοχής και η συζήτηση των τροπολογιών. Ο κύριος Κόλιτσεκ όμως δεν μπόρεσε να παραστεί ούτε κανείς άλλος από τους συνεργάτες του. Άρα, να, διαβάσουμε το κείμενο του κύριου Κόλιτσεκ. Εγώ είμαι μόνο αγγελιοφόρος, οπότε μη με πυροβολείτε. Για όλα τα, τα επίμαχα σημεία τα οποία τυχόν θα αναγύψουν έτσι, λοιπόν, είναι επιστολή επιστολέ μα. Το να σα το διαβάσω. Λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ για τη συμβολή σα. Και επίση σα ευχαριστώ και την γραμματεία για όλα όσα βοήθησε όσον αφορά τη συνεργασία μα. Και από ό,τι καταλάβατε, οι περισσότερε από τι προτάσει μα αφορούν εκείνο το χρήσιμο έγγραφο εργασία τη Επιτροπή. Και επίση είπαμε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα κενά που υπάρχουν για τι δαπάνε, για την πολιτική συνοχή. Θα έπρεπε να υπάρχει συνοχή σε έργα σχετικά με τον σιδηρόδρομο και σε τρόπους μεταφοράς φιλικού στο περιβάλλον και ότι θα έπρεπε με κάθε τρόπο να μειωθούν οι εκπομπές ε, διοξειδίου του άνθρακος. Όσον αφορά δε τις προτάσεις σας, ε, κατάλαβα ότι αυτά τα οποία θέλετε είναι να έχουμε ως αφετηρία της υπόψης της Επιτροπή μας και έτσι να αξιοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου σύμφωνα με τις καθημερινές γραμμάς και πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες. Αποδέχομαι ως προφορική τροπολογία την πρόταση Λιμπεράσκη. Ε, κάτι το οποίο θα αποτελεί μια προσθήκη νέας παραγράφου στο 2α γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο συνάδει με το έγγραφο εργασία μας. Οι τροπολογία 1, 4 και 7 εν μέρει η βαθμό 8, 9, 10, 11, 12 και 19 αυτές ε, όλες νομίζω ότι είναι θετικές όσον αφορά το στόχο και είναι πάρα πολύ θετικά όσον αφορά τις προστεραιότητες, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαφάνεια για τα διάφορα έργα και το ίδιο συναφορά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτά ε, έχουν να κάνουν και με την αποτελεσματική χρήση ενέργεια αλλά και με κάποια ευθύ συστήματα μεταφορών. Προτείνω αποχή όσον αφορά το δεύτερο τμήμα τη 8. Διότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί για κάποιο θεωρητικό σχήμα που μας οδηγεί σε περιπτωσιολογική εξέταση της, ε, της κάθε περίπτωσης 3, 4 και 40 αφορούν κάποια κείμενα με λιγότερες πληροφορίες όμως ε, αντί για αυτές θα ήταν πιο χρήσιμο να κάνουμε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι της Περιφερειακής Επιτροπής Γιατί έτσι είναι δεν έχουμε πιο βιώσιμε επενδύσει για τι μεταφορέ. Οπότε παρακαλώ εδώ πέρα να κρατήσουμε το αρχικό κειμένο και το οποίο εγώ πρότεινα για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι το πιο πρόσφορο για του στόχου μα τώρα όσον αφορά την τροπολογία υπαριθμών 5 και όσον αφορά την εκτέλεση κάποιων προγραμμάτων. Εδώ δεν έχει σχέση με επάρκεια ανεπάρκεια των φόρων, διότι τα κράτη-μέλη εδώ θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε τι οικονομικέ και άλλε διότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω αξιολογήσει, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση των προβλεπόμενων έργων στι επικράτειέ του κατόπιν των όσων προβλέπει ο κανονισμό για την χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων, οι 6, 11 και 16, ε, αυτέ ε, τι τείνουν να είναι περιτές ή ακόμα χειρότερα παραπλανητικέ. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί το ότι θα πρέπει να έχουμε συνδυασμένε μεταφορέ και για το σιδηρόδρομο που να εμπλέκεται και θα πρέπει μεγάλη προσοχή να μην εδώ πέρα εμπλέξουμε κάποια διασυνοριακά προγράμματα που έχουν να κάνουν με τις εθνικές αρμοδιότητες ε, και αυτό που εδώ προτείνεται είναι χρήσιμο αλλά ίσως δεν είναι το πιο δόκιμο στα πλαίσια αυτής της εκθέσεως επίσης προτείνω οι 16 και 18 να απορριφθούν οι 16 διότι είναι θέμα προπολογίζουμε εδώ να δούμε κατά πώς τι θα γίνει όσον αφορά τα λάθη των ε, ε, κρατών μελών και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν τίποτα στοιχεία για τίποτε τέτοια ασφάλματα και ε, για τη δεύτερη το πρόβλημα που σας είπα, διότι εδώ αφορά και τις δημοκρατικές αποφάσεις και διαβούλευση που θα πρέπει να κινούνται σε, κάποιες, με κάποιες δικαιολογίες, ε, διαδικασίες ε, διαφανείς στα πλαίσια των εθνικών νομοθετήτων. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, για την κατανόησή σας. Α, αυτά είναι οι δηλώσεις του κυρίου Κόλιτσεκ όσον αφορά την έκθεσή του. Mr. Κύριε Ιταλά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω να σας πω πρώτα ότι πέτυχε. Ο εισηγητής πέρασε το μήνυμα όσον αφορά για αυτούς τους πόρους από διευθυντικά ταμεία και ταμείο συνοχής που αφορούν τις μεταφορές. Ότι θα πρέπει να με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να ε, ε, αναδειχθούν τα, τα προγράμματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών κλπ. Εγώ πάντως από αυτά που είπατε για τις τροπολογίες που δεν θέλει ο Εσύ συμφωνώ μαζί του για το 18. Επίση, καταλαβαίνω αυτό που θέλω να μα πει τι απόψει του. Και ε, ε, όσον αφορά επίση την τροπολογία υπαριθμών 2, νομίζω ότι δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Είναι θέμα διατύπωση. Όμω, μια που δεν συμφωνήσαμε για τη 2, την αποσύρω. Και συμφωνώ με την 18. Κύριε Σενιαλόβου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λιμπεράτη που τον σχεδόν ηγητή μα δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στι ε, συναντήσει, οπότε να σα πω για κάποιε τροπολογίε τη γνώμη του. Χώρισε το, το υλικό εδώ σε δύο ημίση, πρώτα-πρώτα για τις τροπολογίες, ε, διστάζει να τις αποδεχτεί. Και δεύτερον έχει κάποια άλλη ομάδα τροπολογιών εκεί όπου διαφωνεί. Για να δούμε τώρα η πρώτη ομάδα τροπολογιών. Ας πούμε η τροπολογία υπαριθμών 7, εκεί που αναφέρει κάποια, κάποια προγράμματα μεταφορών, είναι μεγαλοσκελή, αλλά συμφωνεί όσον αφορά την ε, τροπολογία 8 και το δεύτερο τμήμα αυτής εδώ μας αναφέρει για κάποιες ε, υποδομέ μεγάλη ταχύτητα συνδυνούν πρωτεύουσε και μάλλον ε, απίθανο είναι ότι ποτέ θα υπάρξει ένα τέτοιο δίκτυο. Και βέβαια συμφωνούμε με τέτοιου είδου υψηλέ ταχύτητε. Αλλά λέμε ότι μάλλον είναι πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό το οποίο λέει. Τώρα κάτι άλλο υπάρχει στην τροπολογία. Υπάρχει μόνο 10 και αυτή είναι σκελή, αλλά είναι σωστό το ότι παραπέμπει στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί όπου Αναφέρεται και η πράσινη βίβλος. 11 τώρα. Για το 11 δεν νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να καλύψουμε τις οδικές μεταφορές. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Τώρα, για το 16. Για το 16. Εδώ είναι θεμητή αυτή η κριτική όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Μάλλον ατυχώ αυτό αναφέρεται εδώ και όπως ε, είπατε αυτό θα κατέβει ω προφορική τροπολογία. Και άλλωστε ο συγκριτή την αποδέχεται γιατί καλύπτει αυτό που θέλει να πει. Και εκείνος όσον αφορά την ε, δεύτερη ομάδα τροπολογιών εδώ έχουμε κάποιες ε, συστάσεις από τον πλευρά του συγκριτού Πρόκειται για την τροπολογία υπαριθμών 3. Εδώ έχουμε κάποιες κάποια κονδύλια για επενδύσεις διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Θεωρεί ο εισηγητής ότι η τροπολογία υπαριθμών 4 είναι καλύτερη. Καλύτερη και η διατύπωση σε σχέση με την υπαριθμών 3. Επομένω δεν θα επιψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 3. Όσον αφορά δε την 4, εδώ καλύτερα η διατύπωση από το αρχικό κείμενο, εδώ πέρα που συγκρίνονται οδικές μεταφορές και συνδρομικές μεταφορές. Εδώ λέγεται ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες υποδομές συνδρομικέ γιατί αλλιώ έχουμε οδικέ ε, ε, υποδομές. Μετά έχουμε ε, συνδέσμενε μεταφορές, έχουμε δίκτυα ΔΕΔ ε, στο 13 έχουμε το αρχικό κείμενο. Μια χαρά. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ πρέπει να εξασφαλιστούν λέει ε, για τα δίκτυα δε κάποιες, ε, κάποια, κάποια κονδύλια και από ό,τι φαίνεται Ε, είχα ζητήσει το λόγο νωρί, Πρόεδρε. Μην με ξεχάσετε όμω εμένα. Εντάξει, τώρα η σειρά δεν έχει σημασία. Ε, ελπίζω, ε, απλώ ήθελα να μην με ξεχάσετε. Ο σκιώδης συγγητής μας δεν είναι εδώ, οπότε θα αναλάβω εγώ να σας πω τι γίνεται. Δυστυχώ δεν είναι παρόντε πολύ. Θα μείνω στα γενικά. Εμείς ε, ουσιαστικά υποστηρίζουμε όλες τις τάσεις, όλες τις παρατηρήσεις που βασίζονται στο να, να συνδέσουμε με την, ε, ε, τις ευρωπαϊκές μεταφορές με την συνοχή. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρονται σε αυτό το υποστηρίζουμε. Δεν υποστηρίζουμε τη συγκεκριμένη παρατήρηση που ισχύει μόνο για διασυνοριακές μεταφορές ή μόνο για διαλειτουργικότητα θέλουμε, ή μόνο για συγκεκριμένους τομείς. Θέλουμε αυτό να ισχύει για όλους τις, ε, τους τομείς μεταφορών έτσι ώστε να δαπανώνται τα χρήματα με τον πιο εποφελή δυνατό τρόπο. Τα διασυνοριακά προγράμματα έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί συγχρηματοδοτούνται λιγότερο από τα κράτη-μέλη, αλλά χρειαζόμαστε νομίζω όλες τις δυνατότητες που έχουμε, για να, που έχουμε από, την, από τα Ταμεία Συνοχής για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την, ε, τις μεταφορές. Για την τροπολογία 4 θα ήθελα να ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία. Αυτή ε, η ε, αυτή η τροπολογία να πάει μέχρι το Intermodal European Transport και μετά να ψηφίσουμε το όλο κομμάτι χώρια. Γιατί για το πρώτο κομμάτι μέχρι και που σας είπα μπορούμε να συμφωνήσουμε, για το επόμενο όμως δεν μπορούμε. Οπότε θα ήθελα να α, ψηφίσουμε ξεχωριστά. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα και ευχαριστώ τον α, εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, ευχαριστώ. Το θέμα αυτό όντω είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί εδώ μιλούμε για το ότι επιτέλους πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε στοχευμένα τα μέσα που έχουμε. Η τροπολογία ε, λοιπόν που ε, υποβλήθηκε από τους δύο συναδέλφους είναι πολύ σημαντική για τα μέσα από το Διευθυντικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λαμβάνονται πάντα τόσο σοβαρά υπόψη. Μιλώσουμε και για την πιο οικολογική πτυχή της, ε, των μεταφορών και για την απαθρακοποίηση των μεταφορών. Οπότε νομίζω ότι... Μονίμως αναφέρονται οι οδικές μεταφορές. Κάτι που ουσιαστικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που, τις ε, κατασκευάζουν, τις, ε, που κατασκευάζουν τους δρόμους για τις οδικές μεταφορές. Ε, κάτι που δεν νομίζω ότι μπορούμε να το επηρεάσουμε εμείς ιδιαίτερα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους και να τους παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας. Το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία που υποβάλαμε εμείς για να έχουμε μια καλή βάση αξιολόγησης. Και, το, και νομίζω ότι πρέπει να το ξαναζητήσουμε αυτό δηλαδή που έχουμε ζητήσει ήδη ως Κοινοβούλιο από την Κομισιόν στην, στο ψήφισμα της 22ης ε, Απριλίου 2009 για, τα, για συγκεκριμένες πληροφορίες για χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Αυτές οι πληροφορίες δεν έρχονται, δεν υπάρχουν, δεν μας δίδονται. Υπάρχουν ε, τροπολογίες για το ότι α, θα θέλαμε να, χρηματοδοτείται να χρηματοδοτείτε περισσότερο το ένα ή το άλλο. Εντάξει, μπορούμε να δούμε τι είναι λάθος και τι είναι σωστό, αλλά θέλουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι μεγάλη έλλειψη. Και χαίρομαι που το υποστηρίζει και ο εισηγητής. Εμείς ζητούμε αυτές τις πληροφορίες. Γιατί ακριβώς ε, επειδή υπάρχει και αυτό το θέμα λιτότητα στα κράτη-μέλη, υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα μέσα και, τα, και αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τον πιο στοχευμένο τρόπο γιατί μιλούμε για βασικές δαπάνε για την πολιτική μεταφορών. Να μην επικεντρωθούμε μόνο στις μεγάλες συνδέσεις επίσης, γιατί μιλούμε και για ε, μικρότερα κράτη που έχουν μικρότερες συνδέσεις και οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές. Ας μην επικεντρωθούμε λοιπόν μόνο σε μεγάλα προγράμματα. Υπάρχει ε, στην Ιταλία, στην Ιταλία μεταξύ δύο ε, σημείων δεν υπάρχει διεθνέ τρένο, διεθνή σιδηροδρομική σύνδεση. Υπάρχουν μόνο τοπικά τρένα. Και αυτό σημαίνει ότι όταν ένα τρένο είναι τοπικό, σημαίνει ότι σταματάει πάρα πολλέ φορέ και επιμηκύνεται ο χρόνο του ταξιδιού. Και επίση δεν είναι το θέμα μόνο αν υπάρχει υποδομή για να υπάρξει διεθνή ε, σύνδεση, αλλά υπάρχει και το θέμα του πώ χρησιμοποιούμε την υποδομή που υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι σημαντικά. Χαίρομαι που αρκετά από αυτά τα υποστηρίζει ο συνάδελφος Κόλιτσεκ. Και επίση ζητούμε και πάλι τι ε, πληροφορίε από την Κομισιόν, γιατί πραγματικά θα μα διευκόλυνε πάρα πολύ και τη ζωή και την συζήτηση, γιατί πρέπει να συζητούμε επί τη βάση συγκεκριμένων πληροφοριών. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ζέλερ. Ε, Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Μια που ζήσει ο Αγγελεφόρο, παρακαλώ να το διαφημίσεις, να το διαβιβάσεις τη συμφωνία μου. Όμως, σας πείσω την προσοχή ότι άσχετα από το ότι η πολιτική συνοχής θα αναθεωρηθεί Παρ' όλα αυτά, μια που το κείμενο αυτό αφορά και τις μεταφορές, τι θα γίνει, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν την ύφη. Γίνεται, υπάρχει χρηματοδότηση. Αλλά προσοχή στα ποσά. Μην θα δώσουμε αυτά στα κρατη και αυτοί κάνουν του ε, υπολογισμού. Βεβαίω, ε, πέρα πρόκειται περί ανάπτυξη και επομένω θα πρέπει να δούμε το πώς θα βοηθηθεί το δίκτυο των ΔΕΔ, αλλά θα πρέπει να αρθούν τα παραθυρά και τα κενά που στο σύστημα. Δεν νομίζω πάντως ότι μόνο με αυτούς τους πόρους πρόκειται να ολοκληρώσουμε την πορεία μας με το 2020. Γι' αυτό και για το 8 και για το 4 έχω κάποιες, ε, ε κάποιες ε, αμφιβολίες. συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα των σιδηροδρόμων είναι τα έργα κλειδιά και θα πρέπει να έχουν η μέρα του λεόντος σιδηρόδρομοι. Αυτό αφορά και τα διασυνορικά προγράμματα και έργα. 12 και 16 επίσης εδώ αναφέρονται κάποιες επικρίσεις όσον αφορά την έλλειψη ισορροπία σε κάποιες επενδύσεις των κάποιων κρατών μελών. Καλά. Εδώ πέρα θέλουμε να αλλάξουν τροπολογία, εμείς δεν συμφωνούμε. Πάντως, εν μέρει συμφωνούμε και αυτές τροπολογίες Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το κείμενο, όπως είπε και η κυρία Λίχτεμπεργκερ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και η κλίδα χρηματοδότηση στον ΕΡΤΕΡΤΕ. Δεν υπάρχει άλλος ε, ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Και πρόκειται για τα χρήματα τα οποία χρηματοδοτούνται ε, σε περιφερειακό επίπεδο από το Περιφερειακό Ταμείο. Καμιά άλλη επιτροπή δεν έχει τόσα κονδύλια στη διάθεσή της. Υπάρχει μία πρόταση μεταξύ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και των κρατών και των περιφερειών που έχουν έναν ειδικό στόχο και τους δικούς μας στόχους που είναι ευρωπαϊκοί. Πρόκειται λοιπόν για μια ουσιαστική αντίρρηση εδώ. Εγώ δεν έχω... Δεν έχω να πω άλλα γιατί δεν είναι εδώ εισηγητής, αλλά να, να επαναλάβω την προφορική τροπολογία στην τροπολογία 13. Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής η Επιτροπή να θέσει και τα όρια αναλογικότητας στο μέλλον. Στο μέλλον δηλαδή να σκεφτεί η Κομισιόν ε, στα πλαίσια της συνοχής να εισάγει στο μέλλον. Αυτό ως προφορική τροπολογία. Ωραία, θα το δούμε αυτό αύριο. Κύριε Γελασάντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του κυρίου Κόλτσεκ για την παρουσίαση που κάνατε, για την, τις πρότασεις και να σας πω ότι στην τροπολογία 13 μου φαίνεται τέλεια η πρόταση που υποβάλλει. να αυτονομήσουμε τις περιφερειακές πολιτικές από τις πολιτικές μεταφορών. Και εδώ πραγματικά με ακούλπα, δικό μου το φταίξιμο. Θα ήθελα να ρωτήσω στη γνωμοδότηση για τη Σούρε να το ξαναδεί και να μην πετάξει στα σκουπίδια την πρώτη πρόταση της τροπολογίας 8 του κυρίου Κόλιτσεκ. Δηλαδή να παραμείνει τονίζει τη σημασία των μεταφορών προκειμένου να εξασφαλιστεί η εδαφική οικονομία και κοινωνική συνοχή. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε ταυτόχρονα συνολικά την αύξηση όλων των ταμείων. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το κοινωνικό ταμείο απ' έξω. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σίμψον εκ μέρους του κυρίου Κόλιτσεκ αν ε, θα δεχθούμε την τροπολογία του κυρίου Λιμπεράτσκι που είναι περισσότερο μια τροπολογία για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και όχι για μας. Δεν κατάλαβα αυτό το 19% τι είναι, δίκτυα τι είναι. Ανησυχούμε διότι δεν αυξήθηκε το 19% της συνοχής, του Ταμείου Συνοχής ή αναφερόμαστε εδώ μόνο στα δίκτυα. Αναφορά μόνο στα δίκτυα, μα δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτή η προφορική τροπολογία σε αυτή τη γνωμοδότηση. Κυρίως να λάβουμε υπόψη την τροπολογία μου φαίνεται ότι ήταν του κυρίου Νταντέ, όπου λέγεται ότι ανησυχούμε γιατί τα διασυνοριακά σχέδια δεν προχωρούν και καθυστερούν. Αλλιώς δεν βλέπω ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ. Έχουμε αυτή την προφορική τροπολογία του κ. Λιμπεράτης και λέμε να την προστάσουμε ε, ως νέα παράγραφο 2α. Όμω τι προτείνει να απορριφθεί η 16 που λέει εδώ πέρα ότι είναι αρμοδιότητα προπολογισμού. Αυτά έχει προτείνει. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Θα γίνει αύριο ψηφοφορία. Το επόμενο είναι η α, έκθεση σε ένα λόγο για κάποιου είδου διατάξεις που αφορούν κινητήρες. Θα να ευχαριστήσω τους δύο και να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτρια για την συνεργασία. Η κυρίως αρμόδια επιτροπή ήταν η Επιτροπή Περιβάλλοντος και θεωρήθηκε επί, παρόσο πάρα πολύ πολύ έκθεση γιατί αφορούσε βιομηχανία και περιβάλλον. Έχουμε 16 τοπολογίες εδώ, δύο απεσχέτησαν, οπότε μας έχουν απομείνει 14 που πρέπει να ζητηθούν. πηγαίνουν προ την ίδια κατεύθυνση κατά την Έχουμε, έχουμε ομοδοποιήσει σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα-πρώτα, αυτές που αφορούν την καταψήφιση της όλης έκθεσης, αλλά καλύτερα θα το αφήσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να συζητήσουμε εδώ τις πιο τεχνικές τροπολογίες, ιδίω εκείνες οι οποίες αφορούν τους σιδερόμους. Τώρα, το δεύτερο τμήμα αφορά στην αναβάθμιση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά δύο τρόπους. Είτε με αντικατάσταση των πιο βρώμικων των μηχανών και ε, αντικατάσταση με κινητήρες στα 2-3α. Εγώ όμως προτείνω αυτό να γίνει με προφορική τροπολογία. Οπότε κατά τέτοιο τρόπο αυτό να γίνει όσον αφορά αυτά τα τρένα. Και επομένω, όσον αφορά την τροπολογία, να μην πούμε τίποτα άλλο, να αφήσουμε τα υπόλοιπα έξω. Τώρα, ένα άλλο θέμα πολλών τροπολογιών είναι το να απονευρωθεί πρόταση της Κομισιόν και να υπάρξουν σωρό παρεκκλήσεις ε, και να γίνουν η αντικατάσταση κάποιων αρχαιοτέρων ε, κινητήρων, μηχανών. Κάτι γνώμη όλες αυτές τις τροπολογίες δεν θα πρέπει να υποστηριχθούν. Σύμφωνο με την πρώτη πρώτη ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Τώρα, η τρίτη μου τροπολογιών αφορά κάποιους, ε, κάποιες μηχανές, ατομομηχανές, οι οποίες έχουν τεθεί σε εμπορία σχετικά με το σημείο αυτό έχουμε διάφορες τροπολογίες. Μη τον οποίο ότι θα πρέπει να λεφθούν υπόψη οι, οι διορυθμίες των σιωδρόμων του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάποιες από αυτές με βρίσκουν σύμφωνο και θα επέτρεπε στους κατασκευαστές αυτών των ατομικανών να έχουν κάποιο περιθώριο στην κατασκευή. Αυτά όσον αφορά τις εν λόγω 14 τροπολογίες. Ελπίζω τελικά θα περάσει το όλο κείμενο γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά ε, ισορροπημένο και είναι αρκετά ε, δίκαιο και σωστό και για περιβάλλον και για την βιομηχανία. Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι εδώ η Κομισιόν θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν ε, ορισμένες τροπολογίες και αντιτροπολογίες που αφορούν στη συνδυασμένη μεταφορά οδική, οδη, ε, συνδυασμένη μεταφορά οδική, οδική και σιδηροδρομική. Λέμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για το ότοράι. Θα έπρεπε λοιπόν να φτιάξουμε ακόμη ένα κείμενο το οποίο θα αφορά στον ορισμό. Αλλά φαίνεται όμως ε, ότι υπάρχει ένας όρος στα πλαίσια της Επιτροπολογίας στην Κομισιόν το 2010 αποφασίστηκε πρόκειται για ορισμό που τον έχουμε στα κείμενα αλλά αυτό είναι ο επίσημος να μας το επιβεβαιώσει η Κομισιόν. Διότι αν υπάρχει ορισμός, εγώ θα ήθελα... Ε, γιατί θα ήθελα το train set να το ορίσουμε στο κείμενο γιατί μιλάμε. Αυτού του τύπου η διακίνηση αφορά στις ανατολικές χώρες οι οποίες έχουν περισσότερες υποδομές αλλά λιγότερα μέσα για να τις χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, ε, σε αυτή το πλαίσιο θεωρώ ότι είναι χρήσιμη ερώτησή μου. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Ως κοιόδηση εισηγήτρια δεν ε, έχω υποβάλει τροπολογίες γιατί αυτά που έγραψε η κυρία Σενιάλοβα έβρισκαν ε, σύμφωνοι, οπότε δεν υπάρχω, δεν είχα να πω εγώ τίποτα άλλο. Κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν ε, ε, υποβληθεί, εντάξει, μπορώ να τις υποστηρίξω, συγκεκριμένε, κάποιες πιο γενικές επίσης μπορώ να τις υποστηρίξω. Οπότε εγώ είμαι στο πλευρό σας. Στην ομάδα μας εμείς επικεντρωθήκαμε στις εξαιρέσεις για, την, για το Ηνωμένο Βασίλειο. και μάλιστα ασχολήθηκα πολύ μαζί με την Κομισιόν και με διάφορους εμπειρογνώμονες γιατί φαίνεται ότι όντω στην ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι ε, υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να έχουμε αυτές τις εξαιρέσεις Εντάξει, αντί να έχουμε ας πούμε 12 παλιές μηχανές και να, τις πάμε, να το πάμε στις 20 για, τις, για την κατασκευή, εντάξει. Αλλά τώρα να αλλάξουμε το χρονικό όριο, να έχουμε δηλαδή τόσο σημαντικές εξαιρέσεις, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δεχτούμε. Το συζητήσαμε επιμακρών στην ομάδα μας, γιατί αυτό είναι ευρωπαϊκή διάταξη Βέβαια, εγώ τον Πρόεδρο τον σέβομαι απόλυτα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε γιατί ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να επιβαρύνουμε το ευρωπαϊκό σύστημα με τέτοιες ε, κραυγαλαίες εξαιρέσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή τη συγκεκριμένη λοιπόν ανθρωπολογία που αφορά αυτή τη χώρα εγώ δεν μπορώ να τη δεχτώ. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Όπως οι περισσότεροι θα περιμένετε, ούτε εγώ είμαι μεγάλη οπαδός του να αποδυναμώνουμε κι άλλο τις ούτως ή άλλως όχι πολύ φιλόδοξες πολιτικές μας. Για μένα ε, είναι λίγο ντροπή είναι λίγο επίπλαστο να πηγαίνουμε σε διεθνείς διασκέψεις και να μιλούμε για τον πρωτοπόρο ρόλο της Ευρώπης και μετά όταν φτάνουμε στο συγκεκριμένο κάποια κράτη-μέλη να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή να, και να κάνουν κάθε τι που είναι δυνατόν να μην αλλάξει ε, το καθεστώς, ε, εκεί δεν, δεν, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Νομίζω ότι αυτή την πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να την απορρίψουμε μόνο την 6 και τη 16. Μπορώ εγώ να δεχτώ Για τις υπόλοιπες τροπολογίες έχω πρόβλημα. δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποδυναμώσουμε μία, την πολιτική τόσο πολύ ώστε να ωφεληθούν κάποιε χώρε που ούτω ή άλλως ωφελούνται τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να ισχύει κάτι α, σήμερα για κάποιε χώρε και κάτι άλλο να μην, και για άλλε χώρε να μην ισχύει. Δεν προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον και προφανώ δεν ξέρουμε και τι θα γίνει σε 30-40 χρόνια αν συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιε κρεβαλέ εξαιρέσει. Ευχαριστώ. It's simple. είναι απλό. Αν θες να αποτελειώσεις τα εμπορικά τρένα, τότε κοίτα αυτή την περίπτωση της παρέκκλησης. Γιατί είναι μια από πάρα πάρα πολύ μικρή θέση στην αγορά. Προβλήματα με τις διαστάσεις, τις ράγες, ε, το βάρος, πολύ χειρότερα από την Ευρώπη. Οπότε, ε, εδώ λέμε το κατά πόσο θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η μικρή ανάπτυξη που καταφέραμε να πετύχουμε ε, αυτή, αυτή το, το, το, το, κάπως έγειρε η πλάστικα να καταφέρουμε αυτό να, να διατηρηθεί γιατί αν, ισχύει, αν τελικά πρέπει να βγουν αυτές οι μηχανές τέλος πράξη θανάτου για αυτά τα τρένα δύο-τρία χρόνια θα χρειαστούν αντικατάσταση. Γι' αυτό και λέμε ότι χρειάζεται αυτή η παρέκκληση. Έχουμε Έχουμε ξέρει το μηχανέ 30-40 ετών στην Κατρίνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όποιο πει ότι αυτό είναι γελίο, ναι εντάξει θα του πω πάσο, αλλά όμω έτσι είναι πραγματικότητα. Αυτό το οποίο λέει το κείμενο είναι ότι με αυτό του είδου την ε, εξαίρεση θα δοθεί μια παράταση για αυτή την νομοθεσία και έτσι θα γίνει η αντικατάσταση με κάποιε μηχανές που θα είναι δυστυχώ από τον Καναδά, πάντω θα είναι καινούριε και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε τα εμπορικά τρένα. Αλλά αν πούμε ότι δεν θα υπάρχει καμία εξαίρεση, τότε τα εμπορικά τρένα θα έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και όλοι μου λένε ότι θα ήταν πάρα πολύ θετικό να μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ακόμη περισσότερα εμπορικά τρένα. Να, προτεραιότητα. κυρία Σρέντερ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σενιολόβα για την εκθεσή τη και σε ευχαριστώ όλους για τις τροπολογίες να σα πω κάποιε παρατηρήσει όσον αφορά τα όσα άκουσα σήμερα πρώτα απ' όλα όσον αφορά την αντικατάσταση των κινητήρων αυτών των μηχανών και το δεύτερο αφορά αυτές τις τι τις ίδιες ε, κάποια θέματα που αφορούν στο Ηνωμένο Βασίλειο πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την αντικατάσταση αυτών των μηχανών. Δεν είπαμε εμεί τίποτα τέτοιο. Θέλουμε να δούμε τι ευελιξία μπορεί να υπάρχει. Γιατί τώρα ο κλάδο αυτό θα πρέπει να υιοθετήσει φιλόδοξου κανόνε να ξεπεράσει την κρίση. Το θέμα της αντικατάστασης των μηχανών είναι οριζόντιο. Ήδη έχει προβλεφθεί και ε, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη μελέτη αναφερτικού κειμένου. Οπότε θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία για την αντικατάσταση. Αυτό θα πρέπει να γίνει με αντικατάσταση οδηγίας η κυρία Σινιαλόβου το είπε. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα για την αντικατάσταση. Πρώτα απ' όλα για την τεχνολογία 3α. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε ότι επιτάσσει τεχνολογία 3α, να δούμε άλλους τρόπους. Τώρα όσον αφορά τις εξαιρέσεις, το μελετούμε. Και να μην έχουμε αυστηρά κριτήρια δεν, δεν πειράζει. Δεν είναι τόσε πολλέ. Το βλέπουμε από δική μα πλευρά τώρα. Όσον αφορά τι ε, ατομομηχανίε αυτέ, πρώτα-πρώτα έχουμε μια σειρά τροπολογιών που έχουν υποβληθεί όσον αφορά τι ε, μα αυτέ. Ε, έχουμε και αυτό το σχήμα τη ευελιξία. 12 έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ γράφει 40 και 50. Ε, δηλαδή είμαστε ανοιχτοί να δούμε τα στοιχεία. Και επίσης να καταλήξουμε σε κάποια τροπολογία που θα τάσει και κάποια όρια εκπομπών που είπαμε ότι είναι σημαντικό για την προσθέτη του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο είδου ε, περιθώριο ελιγμών. Ο κύριος Ρικέ κάτι συγκεκριμένο είπε όσον αφορά ε, αυτούς τους, αυτά τα μηχανήματα. Έχω μια απόφαση του 2010. Και μέσα από την Επιτροπολογία και είχαμε προσθέσει να έναν ορισμό που θα τόσο για περισσότερους. Καλή πρόταση Κάτι άλλο τώρα το οποίο συζητήθηκε είναι το θα γίνει με τα κρατη που έχουν διαφορετικά προβλήματα υποδομών. Το Μέρο Βασίλειο αναφέρθηκε. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Και ενδεχομένω έχουμε και άλλα ένα-δυο Το οποίο πρόβλημα. Coaching σε σχέση, σχέση με το παγόνι μηχανές. Δεν ε, έχουμε αντίρρηση ότι υπάρχει διαφορά από κράτος σε κράτος. Βεβαίω εμεί πάντοτε προτιμάμε την πλήρη εναρμόνιση. Επίση είμαστε ανοιχτοί. Να το κοιτάξουμε. Η οδηγία δεν αφήσει και μένα κράτο μέλο. Επικαλείται κάποια χρήσιμα κριτήρια. που τα, τα, το μεγέθους των ε, ραγών, των γραμμών, ούτως ώστε να μπορούν αυτές οι αλλαγές να είναι αποδεκτές. Και εμείς εργαζόμαστε και με κοινοβούλιο και με συμβούλιο. Πάνω σε αυτήν την ιδέα πάντως. Ήδη και τέτοιες διατάξεις ε, έχουν περάσει ε, σε πολλά κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Πέρασε η ώρα. Προσπαθούμε τώρα να κλείσουμε με τις τροπολογίες, αλλά... Τι να κάνουμε, τα αφήσουμε όλα αυτά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω και πάρα πολλά να προσθέσω. Να ψηφίσουμε αύριο, πρόεδρος, πάρα πολύ ωραία, αύριο θα γίνει η ψήφιση. Το επόμενο θέμα στη μέση διάταξη είναι οι προκλήσεις για την πολιτική μας και για τους πόρους και τον προπολογισμό για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή το 2013 είναι δική μου αυτή η έκθεση να δούμε το πρώτο κείμενο. Να σας πω συναδελφοί ότι πρόκειται για μία από αυτές τις κλασικές αποφάσεις των συντονιστών. Ο εισηγητής να γράψει την έκθεση και κατόπιν να του φορτώσουμε 48 τροπολογίες τέλος πάντων. Έχω να σας πω κάποια γενικά θέματα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ευσύνοπτη να διακρίνεται από ακρίβεια αυτή η οδηγία και η άποψή μας να ακούγεται όσο γίνεται πιο σαφής. Όχι, εδώ πέρα δεν είναι το θέμα του να πλασάρουμε τις μεταφορές ε, ως ε, ύψιστη τροπεριότητα. Απλώς θα πρέπει να έχουμε ψηλή στο πλαίσιο του προπολογισμού για, για τις μεταφορές. Οπότε αυτά τα συζητάνε στις αρμόδιε επιτροπές. Άρα δεν είναι θέμα το να αναφέρουμε όλα τα που μας βοηθούν ε, για τις μεταφορές. Όμως θα πρέπει να πούμε τι προτεραιότητες θα πρέπει να τεθούν. Αυτό θέλουμε να ξέρουν όλες οι νομικές επιτροπές. Προσπάθησα εδώ να μην είναι ούτε πάρα πολύ γενικό, και ούτε πάρα πολύ συγκεκριμένη αυτή η Επιτροπή. Γιατί έχουμε κάποιε τροπολογίε οι οποίε τονίζουν πόσο σημαντικέ είναι οι μεταφορέ για τη συνοχή. Και επίση εδώ έχουμε και ε, θέματα τη βιομηχανική πολιτική. Έχουμε κάποιε τροπολογίε που είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει προσβασιμότητα στο σύστημα μεταφορά. Υπάρχουν κάτι άλλε τροπολογίε οι οποίε αφορούν την ε, ανάπτυξη εν του 2020 και κάποιες άλλες που τονίζουν ότι οι φορεί και οργανισμοί των μεταφορών θα έχουν όλο και περισσότερε αρμοδιότητε και αλλού αναφέρεται ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Ε, Επίση υπάρχει. Ε, υπάρχει μια τροπολογία για το πολιτεύει δημοσιονομικό πλαίσιο για τις, για τις ε, ε, ρηπαντικές εκπομπές. Άρα προσπάθουμε να καλύψω όσο γίνεται περισσότερα. Επίσης προσπαθούμε εδώ να έχουμε και συμβαστική διατύπωση, παράγραφο 4. Ας πούμε λέμε ότι εδώ θα πρέπει να καλύψουμε το πώς θα είναι ο τομέας των μεταφορών ε, πιο αποτελεσματικός. Είναι πρόκειται για πρόταση κυρίας Γένσεν. Και επίσης θα πρέπει οι πόροι του Ταμείου συνοχή να χρησιμοποιούνται καλύτερα για τις μεταφορές, να ληφθούν επίση οι ευαισθησίε όσον αφορά τι συνεχιζόμενες ε, επαφέ μα με την Περιφερειακή Επιτροπή. Έχουμε και την τροπολογία ΖΙΛ που λέμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί γενικώ η χρηματοδότηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό που δεν ήθελα να κάνω είναι να αρχίσω να ασχολούμαι με το τι είναι καλό και τι είναι κακό για κάθε συγκεκριμένο τρόπο μεταφοράς. Επαναβάλλουμε ότι εδώ πρόκειται για τη συγκεκριμένη ειδική επιτροπή ε, για τις προκλήσεις και θα πρέπει εδώ να δείξουμε ποιες θεωρούμε προτεραιότητες. Άρα εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ότι τα τρένα είναι υπέροχα και τα αυτοκίνητα απέσια. Η πολιτική μας θα πρέπει να είναι να έχουμε ε, ευρύτερα επιχειρήματα για το πώς αυτήν την δική επιτροπή θα την ε, πείσουμε ότι οι μεταφορές είναι η προτεραιότητα. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε. Και οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να δώσουν τη μάχη τους και εμείς τις πολιτικές ομάδες, ώστε να έχουν προτεραιότητα ε, ε, οι μεταφορές με την Επιτροπή Και αυτό το οποίο δεν θέλω να γίνει είναι να αποπροσανατολίσουμε τελείως την Ειδική Επιτροπή για τις προκλήσεις γιατί θα ζητάμε συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα έργα και δεν θα έχουμε μια ευρύτερη άποψη λέγοντάς τους να, ποιος είναι ο λόγος για τους οποίους, αυτή η λόγη για του οποίου θα πρέπει μεταφορές να είναι μια προτεραιότητα. Και ο λόγος ε, αυτός είναι ότι θα πρέπει στα 2020 να, να καλυφθούν αυτές τις προτεραιότητες και όχι να προσαρμόσουμε την πολιτική του 2020 στις προτεραιότητες που θέλουμε. Όλα αυτά προσπάθησα να τα αναφέρω και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να δουλέψουμε και έτσι να προσεγγίσουμε την Ειδική Επιτροπή. Έτσι θα πλασάρουμε τις απόψεις μας. Και να αναγνωριστεί την προτεραιότητα οι μεταφορές. Εγώ αυτή τη συμβολή έχω και ζητεί το λόγο κυρίως Γκρός. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπατε. Εμείς από το ΕΛΚ συμφωνούμε και με αυτό που είπατε για την ε, λίστα της ψηφοφορία συμφωνούμε και με τις περισσότερες ε, τροπολογίες συμφωνούμε. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία δεν μας ικανοποιούν. Σημαντικό για μας είναι οι μεταφορές να ε, λάβουν τη σωστή, συζή... τη σωστή θέση που τους πρέπει στην όλη συζήτηση και για τώρα και για το μέλλον. Θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση με τους πόρους που υπάρχουν για την κινητικότητα. Ούτως ή άλλως ε, στην έκθεση σας αυτό αναφέρεται αρκετά έντονα. Τώρα για το περιβάλλον, για τα οικονομικά, ε, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Ο χώρος των μεταφορών πρέπει να ανοίξει στην Ευρώπη, πρέπει να έχει υγιή ανταγωνισμό, να μην υπάρχει προστατευτισμός ούτε από χώρα ούτε από τομείς. Το, η οικονομία και το περιβάλλον ε, νομίζω ότι μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Δεν χρειάζεται το ένα να αντίκειται στο άλλο. Επίσης όμως πρέπει να, ε, να συνδυάσουμε την πραγματικότητα με τους στόχους μας. Γι' αυτό υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε αρκετούς τομείς. Δεν θέλω να μπω τώρα στη λεπτομέρεια της έκθεσής σας. Ε, συμφωνούμε με πολλά πράγματα. Δεν είναι πολύ λεπτομερής. Μ' αρέσει και το στυλ που έχετε γράψει. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα βέβαια. Πρώτη τροπολογία. Τροπολογία 4. Στο δεύτερο τμήμα, ε, το δεύτερο τμήμα δεν μας ικανοποιεί. Θέλουμε να ολοκληρωθεί, να ολοκληρώνει την τροπολογία στο especially και το υπόλοιπο να διαγραφεί. Άκουσα στην τελευταία, στον τελευταίο κατάλογο υπήρχε μια ε, προφορική τροπολογία για την τροπολογία 1 ε, υπάρχει, εμείς θέλουμε ως ΕΛΚ ξεχωριστή τροπολογία, ε, ξεχωριστή ψηφοφορία, συγγνώμη. Στην 11 θα απέχουμε. Τροπολογία 15 το ίδιο. Στο δεύτερο τμήμα, το δεύτερο τμήμα δεν μας ικανοποιεί, δηλαδή ε, τροπολογία 22 επίσης δεν μας ικανοποιεί. Δεν μπορώ να σας απλουστεύσω περισσότερο τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να σας πω. Α, για την 29 ε, υπάρχει μια προφορική τροπολογία ε, για να υπάρξει καλύτερη Συμβιβαστικές προτάσεις που προτάθηκαν 2, ε, συμβαστική πρόταση 2 δεν έχουμε πρόβλημα. Ε, τροπολογία 13 γίνεται μια μικρή αλλαγή στην τροπολογία της κυρίας Γένσεν. Με την τροπολογία αυτή εμείς συμφωνούμε. Να πω απλώς ότι η τροπολογία 37 στη γερμανική μετάφραση είναι λάθος. Στα αγγλικά λέμε για ε, δάνειο και στα, γερμανικά μιλούν για μισθό. Οπότε καταλαβαίνετε. Απλώς θέλω να πω ότι ε, όταν θα μιλήσουμε για την 37 να ψηφίσουμε την αγγλική εκδοχή του κειμένου και όχι την γερμανική. Εάν το έχω καταλάβει καλά. Ελπίζω να βγάζει νόημα αυτό που λέω. Αυτά πρόεδρε. Ευχαριστώ sure they Ο ε, ehm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Η ομάδα μας ε, συμφωνεί με το σκεπτικό σας και στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα. θέτοντας τις, τις μεταφορές ε, στην καρδιά της συζήτησης και αυτό βέβαια θα γίνει στην Επιτροπή ΣΟΥΡ. Το μήνυμα πρέπει να είναι ότι οι μεταφορές αποτελούν ε, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταφορές ε, θα πρέπει να αποτελούν ένα ενωτικό στοιχείο σε όλες τις πολιτικές και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές στον προπολογισμό για τις μεταφορές και πώς μπορούμε να τις αυξήσουμε. Πρέπει να δούμε τη διαλειτουργικότητα και πώς εμείς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μέσω του Ταμείου Συνοχής για τα σχέδια εκείνα τα οποία έχουν ευρωπαϊκή υπεραξία. Το ίδιο ισχύει και για τα δίκτυα. Περισσότερο από ό,τι σήμερα στο μέλλον θα πρέπει να παλέψουμε για τις διασυνοριακές μεταφορές και τον καλύτερο συντονισμό. Αν εμείς θα πάρουμε όλα αυτά τα μηνύματα και τα περάσουμε, θα έχουμε εκπληρώσει μέγα μέρος των ονείρων μας περί μεταφορών. Αλλά βέβαια θα μας συνεζητούν συνέχεια μεγαλύτερες προσπάθειες. Και οι πολιτικές μας ομάδες και το Κοινοβούλιο. Κυρία Γιάνσεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εμείς ορισμένοι ε, τόσο από εμά και ο κύριος Ρικέ δουλεύουμε στην Ειδική Επιτροπή και επομένω, θα δώσουμε και τη μάχη για το θέμα των μεταφορών. Πάρα πολύ καλά τα λες, Πρόεδρε. Και συμφωνώ. Πώς θα να πω ότι ίσως δεν χρειαζόμαστε τέτοιες συνοριακές ρυθμίσεις, αλλά Ίσως θα πρέπει να τονίσουμε αυτό τις συνδυασμένες μεταφορές για να έχουμε την αποτελεσματική χρήση ενέργειας. Εδώ, εδώ έχουν σημασία οι συνδυασμένες μεταφορές και συγκεκριμένα κέντρα μεταφορών τα οποία θα πρέπει να στηθούν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πολύ σημαντικό είναι αυτό το σημείο. Πάντως, Συμφωνώ. Και ευχαριστώ που, που λαμβάνει υπόψη κάποιε δικέ μου τροπολογίε. Να βλέπω εδώ πέρα και για την ε, ε τροπολογία Τικάου, για τον Γαλιλαίο. να λάβουμε υπόψη κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές. Καλά δεν λέω βέβαια να, πω, να τα πούμε συγκεκριμένα, αλλά και με συγκεκριμένα νούμερα. Είναι μάλλον αυτό πρόημο. Όμως να δούμε τι γίνεται διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. Να μην κατηγορήσουμε τον ένα τρόπο μεταφοράς και τον άλλο. αλλά να δώσουμε μια εικόνα τώρα και τελευταία. Έχω εγώ μια τροπολογία για το Μαρκοπόλο. Λέω ότι είμαι καψηφυλακτική, γιατί λέω ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις εγγυήσει του προγράμματος Μαρκοπόλο Και έτσι ίσως θα μπορούσαμε να λύσουμε κάποια τα προβλήματα. Μην είναι ένα γραφειοκρατικό πρόγραμμα. Όποιο τα πάει καλά θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα και όποιο δεν τα πάει καλά επίση το ίδιο. Μήπω μέσω των εγγύσεων βρεθεί μια καλύτερη λύση. Γενικά συμφωνώ με την γραμμή σου, Πρόεδρε και να δούμε για ποια θα είναι τύχη της τροπολογίας Πολύ καλά λέει ο Κυρία Ντυρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σύντομα. με την άποψή σας να προχωρήσουμε κατευθείαν στο ψητό χωρίς να διαχειόμαστε. Λοιπόν, τέσσερις τροπολογίες. Πρώτη, όχι μόνο, δεν πρέπει να πιστούμε μόνο τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακος αλλά και τη μείωση των δυστυχημάτων, την ε, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ. Δεύτερη τροπολογία. Η εν, εναλλαγή του εξωτερικού κόστους των μεταφορών. Και θέλω να πω και στους συναδέλφους ε, που όπως και εγώ είμαστε στην Επιτροπή ΣΟΥΡ για να εξισορροπήσουμε το εξωτερικό κόστος θα πρέπει να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, δηλαδή χωροταξική πολιτική, συνοχή, δίκτυα μεταφορών, ε, θέματα υπαίθρου, χωροταξικά αστικά θέματα κλπ για να έχουμε πιο αποτελεσματικές μεταφορές. Τροπολογία 21 για το θέμα του εξυγχρονισμού του στόλου. Αν έχουμε έναν καλύτερο σιδηροδρομικό στόλο και κυρίως ε, για θέματα εκπομπών θορύβου, τότε δεν χρειάζεται να χτίζουμε και τους ε, τείχους ε, κατά του θορύβου. Και τελευταία τροπολογία αφορά τα μικροσχέδια μπορούμε να υποστηρίξουμε όπως το προάσπισε και ο συνάδελφος για τον τουρισμό μπορούμε εμεί ε, να υπερασπιστούμε μικροσχέδια τα οποία υπόσχονται όμως πολλά για το μέλλον αντί να έχουμε εμείς μακρόπνοα σχέδια με μελλοντολογική απόδοση. Θα έπρεπε λοιπόν να μην διαχυθούμε, θα έπρεπε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στον τομέα των μεταφορών. Κύριο Ζήλερ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την δουλειά που κάνατε. Για κοιτάξτε λίγο την παραγραφό 9. Εκεί συζητήσαμε και μία δική μου πρόταση και κάτι άλλες. Και κατέληξαμε σε κάτι σαν συμβασμό. Ίσως θα πρέπει να δούμε εδώ και την υπαριθμόν 28. Να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε και εκείνον όσον αφορά την συγκέντρωση του, της εθνικής χρηματοδότησης και αυτά τα δίκτυα. Πώς μπορούμε να συνδυαστούν λοιπόν αυτές τις δύο τροπολογίες. Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος διότι χάρη του, του Προέδρου με ενέπνευσε και θα αποσύρω και την τροπολογία μου 24. Η κυρία Τικάου. Πρόεδρε ευχαριστώ. Στα Ρωμάνικα. Συγχαρητήρια για την έκθεση. Νομίζω ότι με αυτή την έκθεση δεν θα πρέπει να τονίσουμε μόνο πόσο σημαντικέ είναι οι μεταφορέ, για κοινωνική, για κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, έτσι θα πρέπει να προσφέρουμε και επιχειρήματα στην Ειδική Επιτροπή για τι προκλήσει, ούτω ώστε να θεωρήσει με υψηλότερη προτεραιότητα τι ε, μεταφορέ και να χρηματοδοτήσουν τα έργα και προγράμματα. Και υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό με τη μετάφραση. De Είπαμε ότι έχουμε εδώ πέρα κάποια σημαντικά στοιχεία για τις ευφύες μεταφορές και είπαμε ότι οι υποδομές χρειάζονται για τα ηλεκτρικά δίκτυα, για τα ηλεκτρικά οχήματα, το GNS, τον ε, Γαλιλαίο και λέω στους συναδέλφους ότι εγώ απέσυρα την τροπολογία υπαριθμών 40 εκεί όπου έλεγα για κάποια συγκεκριμένα ποσά χρηματος για το GNSS. Εδώ και καιρό αυτό το έχω γνωστοποιήσει και σας επαναλαμβάνω. Πρόκειται για τροπολογία παριθμών 40 την οποία και απέσυρα. Εδώ προβλεπόταν συγκεκριμένα ποσά. Την απέσυρα διότι θεώρησα ότι τα θέματα αυτά καλύπτονται από άλλες τροπολογίες. Εκεί που ζητούνται, δηλαδή περισσότερα χρήματα για το GNSS. Ευχαριστούμε πολύ, κύριος Κράμερ. Σωστό είναι που στην στρατηγική 2020 συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές. 30% των εκπομπών προκαλούνται από, ε, διεξουδίου του άνθρακα προκαλούνται από τον τομέα ε, των μεταφορών, περισσότερο από, από άλλους τομείς. Ε, μιλούμε για μείωση παρόλα που μάλλον προβλέπεται αύξηση στο 35%. Οπότε είναι καλό που το έχουμε αυτό στην ε, πολιτική για το 2020. Ε, σε, για δύο τροπολογίες θέλω να πω κάτι. Τροπολογία 21. Ο εισηγητής λέει στην αρχή ότι θέλουμε να μπούμε στη λεπτομέρεια και να συνδέσουμε τις λεπτομέρειες με τις γενικές αρχές. Ναι, αλλά για το θόρυβο μόνο στις υποδομές υπάρχει συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση του θορύβου. Στο ERTMS το έχουμε δει. Οι συνέπειες δεν έχουν να κάνουν όμως μόνο με τις, με τις υποδομές, αλλά και για, και με τον εξοπλισμό. Στον, ε, στο, για το θόρυβο όμως μπορούμε να δαπανίσουμε πολλά χρήματα μειώνοντας πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά ε, το θόρυβο εάν επενδύσουμε στον εξοπλισμό. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί ο εισηγητής το 2021 αρνείται αυτό, γιατί αυτό ακριβώς που έχει καταγραφεί κιόλα είναι ο λόγος που, ή μάλλον είναι ο τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε το θόρυβο. Νομίζω λοιπόν ότι ο εισηγητής θα πρέπει να το ξανασκεφτεί είναι σημαντικό. Θα έχουμε μεγάλα πλεονεκτήματα. Αν μπορέσουμε να, να διαχειριστούμε το θέμα του, της συγχωρήπανσης, νομίζω ότι θα έχουμε σημαντικές, σημαντικά πλεονεκτήματα για τον τομέα των σιδηροδρόμων. Τώρα, για την μετάφραση. αναφέρονται τα φορτηγά στο, στην θέματα της συγχωρήπανσης. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένο όρο στη γερμανική τουλάχιστον μετάφραση. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά δεν μιλούμε για φορτηγά, μιλούμε για ε, καμιόνια, για τους σιδηροδρόμους που μεταφέρουν για εμπορικά τρένα ουσιαστικά μιλάμε. Δεν μιλούμε για φορτηγά. Θέλουμε ούτω ή άλλω το φορτίο και οι μεταφορές από, τον, από τα φορτηγά να περάσουν στο σιδηρόδρομο. Ε, τροπολογία 34 τώρα. Τι ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε τα, τις συνέπειες με τα λιγότερα δυνατά χρήματα και με τον καλύτερο ε, δυνατό τρόπο να τις διαχειριστούμε. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, χρειαζόμαστε καλύτερη πολιτική. Εάν ε, τηρήσουμε τα μεγάλα προγράμματα, είναι το ίδιο κάνει αν θα είναι τα προγράμματα αυτά έτοιμα σε 10-20 χρόνια κατά 50-30 ή 60%. Αλλά μιλούμε για την καλύτερη διαχείριση. Στην πολιτική μεταφορών μπορούμε να κοιτάμε τα άστρα και για τους επόμενους για τρεις-τέσσερις αιώνες αν θέλετε. Αλλά αν δεν κάνουμε τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση να το διαχειριστούμε το τομέα αυτό. Ε, ευχαριστώ. να συγχαρώ εγώ και για την έκθεση αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει το θέμα. Σχετικά με τα διάφορα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ώστε να παλέψουμε το θέμα στην ΣΟΥΡΕ, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Περιφερειακή. για να μην ε, χάσουμε πραγματικά όπως ε, χάσαμε πέρυσι στις ε, δημοσιονομικές προπτικές όπου εντάξει κέρδισε η έρευνα που είναι σημαντική για την Ευρώπη του 2020 αλλά... τώρα δεν θα πρέπει να μας ξεφύγουν οι υποδομές πόσο μάλλον οι υποδομές ε, για την ηλεκτρική ενέργεια. Θα... <coughs> Δεν θα έπρεπε λοιπόν να χάσουμε και για μια ακόμη φορά αυτό το τρένο όταν έχουμε υπόψη μας και τον ανταγωνισμό της Κίνας και της Ινδίας αυτούς τους τομείς. Χαίρομαι που δεχτήκατε τις τροπολογίες που πρότεινα, διότι όπως είπε και ο κύριος Γκρός, η πολιτική μεταφορών θα πρέπει να χρησιμεύσει για να μειώσουμε και το θέμα των εκπομπών αλλά και να διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που αποσύρετε και την τροπολογία 9 διότι ε, δεν βελτιώνει την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κομισιόν, ο κύριος Ρόιτερς. Πρόεδρε, εξωτιμοί βουλευτές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο το οποίο επιτελέσατε για αυτήν την άριστη νομοδότηση η οποία συνάδει προς τους δικούς μας στόχους, βοηθάει το δικό μας έργο και βεβαίως έτσι καλύπτονται και τα δικά μας ε, δικά μας στόχη όσον αφορά την προσβασιμότητα, την στατική για την ανάπτυξη, τη συνοχή και για τη διαλειτουργικότητα. Αυτό το οποίο έχουμε πει και εμείς στο κείμενο μας και τώρα. Εάν κανείς θέλει κάποιες τροπολογίες που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, αυτό σίγουρα θα αφαιρέσει το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς την Επιτροπή Σούρα. Γιατί αυτό το οποίο θέλετε είναι άλλο, είναι να είναι ψηλά στην προτεραιότητα οι μεταφορές, πολιτικών μεταφορών και οπότε. Πάρα πολλά τα είπες πρώτα στην αρχή, στην εισηγησή σου και σε ευχαριστώ για τη συμφωνία μαζί μας. Και επίσης περιμένω πώς και πώς, πώς να συνεργαστούμε στο μέλλον μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρώτος συνάδελφος σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσει σας. Ξέρω ότι με το που δεν συμφωνούν και αυτές θα θεωρούν ότι προσδίδω εισαγωγικά κάποια θέματα των μεταφορών. Όμως δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να είναι πολιτική αυτή η, η έκθεση και όχι έκθεση για τις μεταφορές. Λοιπόν, δεν θέλω να το με λεπτομέρειε στη Σούρα. Θέλω να αναλυθούμε κάποια βασικά θέματα. Και εκεί θέλουμε να εστιαστεί η προσοχή μας. Γι' αυτό και όντω ήμουν κάθετο σε διάφορα σημεία και είχαμε και κάποιε τροπολογίε. Κύριε Ζήλε, κάτι είπατε για τη συγκεκριμένη σα τροπολογία ή την τροπολογία του κυρίου Μπαλσάιδη, δηλαδή την 28. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την 28, ούτε και με την 33 ε, που επίσης είναι του κυρίου Μπαλσάιδης. Κάπου λέγει για περιφέρειες και εκεί είπε ότι αυτό δεν μ' αρέσει. Λέτε δύο βασικοί χρηματοδότες για τα ΔΕΔ είναι οι περιφέρειες όμως. Αυτό ισχύει για κάποια κρατημέλη, όχι σε όλα. Δεν έχουν να όλοι οι περιφέρειες για κάποια κρατημέλη. Ας πούμε στο δικό μου κράτος μέλος. Και γι' αυτό και ήμουν κατά αυτού του σημείου. Ένα άλλο τώρα. Ένα άλλο σημείο το οποίο ήταν ανακριβές και γι' αυτό επίσης υπάρχει σε εκείνο και οπότε γι' αυτό και προσπάθησα εδώ να τα συνδυάσω. Και με την κυρία Γιάννη μπορούσαμε να βρούμε κάποια διατύπωση. Και με το μάθημα για τη δική τροπολογία. Καλά, να δούμε τι θα προκύψει αύριο. Όχι, δεν είναι καθόλου προσωπικό. Ιδίω αφού ό,τι έγινε, έγινε από τους συντονιστές. αυτό το οποίο θέλουμε είναι οι μεταφορέ να είναι υψηλή προτεραιότητα. Αυτό ψάχνουμε να κάνουμε. Μάικλ, θες το λόγο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε, σαν είναι δυνατόν, και η χρηματοδότηση να αφορά το τροχαίο υλικό και όχι μόνο τις Και έτσι ισχύει γενικά. because I'm not so sure in certain... Πρόεδρος, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει σε κάποια μέλη όπου για παράδειγμα έχετε κάποιους ιδιωτικούς σιδηροδρόμους. Θα, θα γίνει κάτι τέτοιο. Καλά, όταν είναι κρατική σιδηρόδρομοι, ίσως ισχύει αυτό που λες. Αλλά, μα και έργα υποδομής κάνουν οι ιδιώτες, το ίδιο είναι. Πρόεδρος, ναι, αλλά συνήθως με κάποιο τρόπο αυτό γίνεται σε κρατικό επίπεδο. Γι' αυτό και επιφυλάσσουν. Καλά, τέλος πάντων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε. Και τώρα έχουν συνεδρία σε συντονιστές. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα και τώρα πάμε στου συντονιστέ.